Good morning. Καλημέρα σας. Ξέρω ότι είναι αρκετά νωρίς. Θα πρέπει όμως να ξαναρχίσουμε την ακρόασή μας που διακόψαμε χθες. Έχουμε τον Επίτροπο Λάσλο Άντορ μαζί μας, είναι ο πρώτος ομιλητής. Είχαμε τα δύο πρώτα τμήματα της ακρόασης για την ενσωμάτωση των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκπροσώπους από ΜΚΟ, από το Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κτλ. Και τώρα, μετά από τα δύο δηλαδή αυτά πρώτα πάνελ, έχουμε δύο άλλα πάνελ από τις 9 στις 11 και το πρώτο πάνελ, φυσικά ξεκινάμε τον κύριο Άντορ, τον κύριο Ιβάνοφ, τον κύριο Σικουλένα και τον κύριο Ιβανόφ. Θα δώσω πρώτα το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο Άντορ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους, κυρίε και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι και πάλι μαζί σας και να αναφερθώ στο θέμα της ε, ενσωμάτωσης των Ρωμά είναι ουσιαστικά μια συμπληρωματική παρουσίαση αυτής που σας έκανε ήδη η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ. Η πρώτη φορά που ήρθα ενώπιον της Επιτροπής σας, 29 Σεπτεμβρίου, σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Απασχόλησης, ήδη μπορέσαμε να έχουμε μια συζήτηση σε βάθος για τα θέματα αυτά. Και είναι σαφές ότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται στην ημέρησια διάταξη και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και επομένω δεν φαντάζομαι την τελευταία τέτοια συνάντηση στην οποία θα εξετάσουμε αυτό το θέμα. Να κάνω καταρχήν μια επισκόπηση της κατάστασης όσο <laughs> έχει. Θυμόσαστε ότι στις 7 Απριλίου του 2010 η Κομισιόν διέγραψε μια πλήρη στρατηγική προσέγγιση στην ανακοίνωσή της για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρωμά στην Ευρώπη έλεγε, έδινε τότε βασικέ προτεραιότητε η ανακοίνωση αυτή για τη δράση τη Κομισιόν και των κρατών μελών σε ένα ευρυφάσμα τομέων που είναι ενδιαφέροντε για την ενσωμάτωση των Ρωμά. <clears throat> Ω γνωρίζουμε όλοι, είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρωμά και κατά πάσα πιθανότητα είναι η πιο κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα και αντιμετωπίζουν ένα σύνολο από πολύπλοκα αλληλένδετα μεταξύ του προβλήματα. Έχουν λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση και εμεί έχουμε μια μεγάλη πρόκληση ενώπιόν μας που είναι μεγάλη και πολύπλοκη. Κατά την άποψή μου πρέπει να υπάρξει δράση τρεις κέριους τομείς. Καταρχήν να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα της, του αποκλεισμού του Ρωμά με συντονισμένες πολιτικές σε διάφορες τομείς. Δεύτερον, να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση και τρίτον, να υπάρχει καλύτερη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις. Θα ήθελα τώρα να αντιμετωπίσω τα τρία, τους τρεις αυτούς τομείς. Ξεκινώ με τις αιτίες του προβλήματος. Πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές που οδηγούν σε μια μειονεκτική κοινωνική κατάσταση για τους Ρωμά στην Ευρώπη. Και πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του προβλήματος, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσουμε την παιδεία για τους νεαρούς Ρώμα, για τα παιδιά των Ρωμά. Αυτό που θα ξεκινήσει το νωρίτερο δυνατό για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν μια ευκαιρία να ξεκινήσουν σε ισοδίκαιο επίπεδο στην ζωή του. Αυτό σημαίνει όχι μονάχα συμμετοχή σε δημοτικά σχολεία, αλλά και στα νηπιαγωγεία. Για να αυξήσουμε τη δυνατότητα απασχόλησης των Ρωμά, θα πρέπει να βελτιώσουμε και την παιδεία τους. Τώρα έχουμε σχολεία τα οποία δεν είναι χωριστά για τους Ρωμά και νηπιαγωγεία που έρχονται σε επαφή και με τα άλλα παιδιά είναι απαραίτητο για να έχουν τη δυνατότητα πλήρου συμμετοχή στην κοινωνία αργότερα. Ο δεύτερο λόγο ε, του αποκλεισμού είναι ο φαύλο κύκλο τη ε, μεταφορά μεταφοράς από την κάθε γενιά στι επόμενες. Χρειαζόμαστε στρατηγικέ οι οποίε θα εξασφαλίσουν την έξοδο από την ένδυα μέσω της απασχόληση. Πρέπει να έχουμε εδαφικέ στρατηγικέ για να προωθήσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση στο Ρωμά, να δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε όπω είναι η παιδεία, οι υγειονομικέ υπηρεσίε και φυσικά και να αυξήσουμε την παρουσία του στην αγορά εργασία. Όταν μιλάμε για την αγορά εργασία, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι τα προγράμματα θα πρέπει να δώσουν και θέσει εργασία για άτομα χωρί ιδιαίτερα προσόντα, γιατί προ το παρόν θα είναι δύσκολο να κάνουμε σημαντικέ αλλαγέ σε αυτή την κατάσταση. Η αντιμετώπιση τη <clears throat> ένδυα είναι κάτι το οποίο έχει υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι το έτος αντιμετώπισης της ένδυας και της ε, κοινωνικού αποκλεισμού. Και επομένω είναι σημαντικό να παίξουμε ρόλο και στρατηγικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν την ανάγκη να, να υποστηριχθεί και το τοπικό και το εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων σε όλους τους τομείς. Εμείς δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, το ευρωπαϊκό αυτό έτος έχει δώσει μια σημαντική πολιτική όθηση στον αγώνα κατά της ένδυας. Καθώς πλησιάζει το τέλος του το έτος αυτό, το ευρωπαϊκό έτος κατά της ένδυας, θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τις ενέργειες αυτές. Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσω της πλατφόρμας κατά της ένδυας και, και του κοινωνικού αποκλεισμού που θα παρουσιάσει αργότερα η Κομισιόν αυτό το μήνα και που είναι ένα σημαντικό εγχείρημα στη στρατηγική του 2020. Η πλατφόρμα αυτή θέλει να υποστηρίξει το στόχο να φύγουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι από τον χώρο τη ένδυα μέχρι το 2020. Θα τονίσει και πάλι τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ορατά αποτελέσματα και να φτιάξει μια πιο δίκαια και περιεκτική κοινωνία Σημαίνει επίσης και μια δέσμευση να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο τα μέσα και τις μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και του Ρώμα. Υπογραμμίζει την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε την κοινωνική ενσωμάτωση, ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσω σε λίγα λεπτά. Επίσης η πλατφόρμα θέλει να εξασφαλίσει μια πλήρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση και εμεί θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ενσωμάτωση αυτών των θεμάτων και σε άλλους τομείς πολιτικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό λόγω των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ομάδες όπως η Ρωμά. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα, <clears throat> σε ένα δεύτερο θέμα που είναι η αύξηση της συνειδητοποίησης, όπως είπα στην εισαγωγή. Εξακολουθεί να είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα στην ενόψη της μελλοντική μας στρατηγικής η κοινωνική ενσωμάτωση των μειονεκτητούσων ομάδων, κατά την άποψή μου, μπορεί να γίνει μονάχα εάν υπάρχει κατανόηση και δέσμευση προς τούτο των κοινωνιών υποδοχής. Η Κομισιόν έχει οργανώσει γεγονότα υψηλής, υψηλού προφίλ στα κράτη-μέλη με μεγάλη παρουσία Ρωμά για να μπορέσει να ενθαρρύνει την ε, καλύτερη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ουγγαρία αυτό οδήγησε σε επικοδομητικό διάλογο μεταξύ εθνικών αρχών και των κοινοτήτων Ρωμά υπό τις αιγίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από αυτό το θετικό παράδειγμα θα λάβει χώρα μια δεύτερη σειρά γεγονότων υψηλού προφίλ στη Ρουμανία τον Οκτώβριο. Μάλλον έγινε τον Οκτώβριο με 500 συμμετέχοντες από όλους τους χώρους της ζωής και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για κοινή δράση των δημοσίων αρχών σε όλα τα επίπεδα μαζί με τις ευρωπαϊκές αρχές και τις τοπικές αρχές και ζήτησαν από τις αρχές αυτές και στις ε, ομάδες στο Ρώμα να εμπλακούν σε ένα διάλογο για την καλύτερη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος άλλων εμπλεκομένων, όπως η ΜΚΟ, επίσης ήταν πολύ σημαντικός. Εμείς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία με το να φέρνουμε σε επαφή όλες αυτές τις, ε, όλους αυτούς τους φορείς σε τακταχρονικά διαστήματα και θα έχουμε και αντίστοιχα γεγονότα αυτού του είδους στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία. Έρχομαι τώρα στο τρίτο σημείο, το οποίο είναι η βέλτιστη χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική συμπερίληψη και ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ρώμα. Η διαφθορτική πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό μοχλό για να υποστηρίξουμε τι εθνικέ προσπάθειε για τη βελτίωση τη κατάσταση των Ρώμα. Το 1 έκτο των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δηλαδή πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν σε στόχο να προωθήσουν την κοινωνική συμπερίληψη μειονεκτικών ομάδων όπω είναι η Ρωμά. Χαιρόμαστε που όλα τα κράτη-μέλη ήδη χρησιμοποιούν αυτά τα ποσά για να υποστηρίξουν του Ρωμά. Πρέπει όμω να αποδεχτούμε ότι πολλές φορές δεν χρησιμοποιούνται πλήρως ή με τον πιο αποδοτικό τρόπο <clears throat> και χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν έχει δημιουργήσει μια δύναμη κρούσης για τους ε, Ρωμά, η οποία θα κάνει μια επισκόπηση της χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενσωμάτωση των Ρωμά και θα προτείνει λύσεις για μελλοντικέ πρόοδους. Όπως ε, μάλλον σας είπε η, πρόεδρος, η αντιπρόεδρος Ρέντινγκ χθε, εμείς εξετάζουμε τώρα τις ε, απαντήσεις των 100 μελών στα ερωτηματολόγια τα οποία τους εστάλησαν. Και η Task Force, η δυναμικρούση, θα κάνει μια έκθεση αφού τελειώσει αυτή η αξιολόγηση. <clears throat> Έντιμα μέλη. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στα επόμενα βήματα στα οποία θα προβούμε. Τον Απρίλιο του 2011 η Κομισιόν θα παρουσιάσει μία νέα ανακοίνωση επί τη βάση της έκθεσης της δύναμης ε, κρούσης θα περιέχει προτάσεις για τη πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην τονή και στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Για το παρόν, η Κομισιόν θα μπορεί να προσκαλέσει τα πιο εμπλεκόμενα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στο φως των νέων πολιτικών για της Ρωμά. Η στρατηγική μας επίσης περιλαμβάνει και την το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι εθνικέ στρατηγικές για τους Ρωμά. Εδώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικέ και ευρωπαϊκέ προσπάθειε την χάνουν πιο αποτελεσματική παρακολούθηση. Θα προσκαλέσουμε τα κράτη να μα παρουσιάσουν εθνικέ στρατηγικές για τη συμπερίληψη των Ρώμα που μπορούν να είναι και τμήμα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμιση. Προετοιμάσουμε του διαχρονικούς πόρου για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013 και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να εστιάσει τι προσπάθειέ του στην υποστήριξη των στόχων τη Ευρώπη 2020, δηλαδή βελτίωση των δεξιοτήτων, των προσόντων, τη κινητικότητα, τη προσαρμοστικότητα και τη συμμετοχή στην κοινωνία και με ιδιαίτερη έμφαση στι μειονότητες όπω η Ρώμα. Στα συμπεράσματα τη πέμπτη έκθεση για τη συνοχή μαζί με τον Επίτροπο Χάν υποστήριξαμε την ανάγκη για διαθωτικοί πόροι να εστιάσουν σε ένα μικρότερο αριθμό κέριων προτεραιοτήτων ιδίω την κοινωνική συμπερίληψη και τη μείωση τη ένδυα. Το Κοινωνικό Ταμείο λοιπόν θα δαπανίσει περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της τρέχουσα περίοδου προγραμματισμού. Αλλά ακόμα και αυτό το ποσό δεν είναι επαρκές και εξάλλου δεν είναι θέμα χρηματικών ποσών, είναι θέμα καλύτερης συνεργασίας και καλύτερης χρήσης μεταξύ των πόρων που υπάρχουν, καλύτερη σχεδίαση, καλύτερες προϋποθέσεις και καλύτερα στοχευμένες παρεμβάσεις. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας με την βοήθεια και των χρηματαγορών να δημιουργήσουν θέσεις και να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης και να μειώσουμε την ε, ένδυα. Εν κατακλείδη, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να τονίσω ότι το θέμα αυτό τη συμπερίληψη των Ρωμά θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην για διαταξή μα. Είναι μια κοινή ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και των κρατών μελών. Η επιτυχημένη κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση στο Ρωμά μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συνεχή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων των Ευρωπαϊκών Φορέων, των κρατών μελών και των διεθνών οργανισμών. Και φυσικά και των φορέων των ίδιων των Ρώμα πρόκειται για ένα σύμπλεγμα προβλημάτων που είναι πολύπλοκο και έχει πολλές αλληλένδετες πτυχές. Πιστεύω όμως ότι δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να το αντιμετωπίσουμε λόγω της πολυπλοκότητός του. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της πιο αποκλεισμένη και της πιο μειονεκτικής μειονότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, for your presentation. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πραγματικά ελπίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο καμπής. Και εκτιμώ ε, τις προσπάθειές σας καθώς και τις προσπάθειες της Επιτρόπου Reading. Ελπίζουμε πως αυτή η έκθεση που βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα αποτελέσει ένα γόνιμο έδαφος για να έχουμε αποτελεσματικό διάλογο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίασή σας και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ανρί Σικλούνα που προέρχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι υπεύθυνο συντονιστή για θέματα Ρωμά να μας κάνει την εισήγησή του. Έχετε το λόγο. Thank you, A colleague of mine who recently visited a Roma settlement. Ένας ε, συνάδελφός μου που πρόσφατα επισκέφθηκε ε, καταβλισμούς Ρωμά στην Βόρεια Ευρώπη μου είπε πως είχε πέρασε άϊπνες νύχτες λόγω του σοκ που έπαθε. Εγώ επισκέφθηκα τους καταβλισμούς πριν από λίγες, ε, λίγα χρόνια και δεν είναι από τους χειρότερους που έχω εδώ. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ε, η απόγνωση ενός ε, απλού Ευρωπαίου πολίτη όταν ανακαλύπτει πως υπάρχει τέτοιου είδους φτώχεια στη μέση της Ευρώπης και εξακολουθεί να υπάρχει παρά από τις δεκαετίες προσπαθειών διεθνών οργανισμών και πολυάριθμων ενώσεων των Ρωμά. Ζητώ συγγνώμη που ξεκινώ με τέτοια απεσιόδοξη αναφορά, αλλά τη μια διάσκεψη μετά την άλλη διαρωτώ με για πόσο καιρό οι χιλιάδες Ρωμά θα εξακολουθήσουν να ζουν σε τέτοιες ε, καταστάσεις, τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε χωριστά σχολεία, να μην βρίσκουν δουλειά και να δέχονται διαρκώς ε, επιθέσεις. Ε, οι δράσεις που κάνουμε έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ριζώνουν. Πολύ ρωτάμε αυτά τα ερωτήματα και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις. Η κυρία Γιάροκα έχει θέσει αυτά τα ερωτήματα όταν λέει στην έκθεσή του ότι παρά την ύπαρξη πολλών μηχανισμών συνεργασία και διαφόρων οργανισμών, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αφορούν την ε, κοινωνική ένταξη των Ρωμά δεν έχουν ε, αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και άρα η επιλογή του να παραμείνουμε στην ίδια πορεία δεν μπορεί να σταθεί. Ίσως θα πρέπει να πούμε δεν θα πρέπει να λέμε ε, ότι όλες οι προσπάθειες ε, δεν απέφεραν καρπούς. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα όμως. Καθώς είπε ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ανθρώπινα δικαιώματα, ο κύριο Χάμεσμι, οι αλλαγές είναι πολύ πολύ αργές και διαρκώς ε, παρεμποδίζονται από εκδιώξεις, καταδικάσεις, ακόμα και σωματικές επιθέσεις. Γι' αυτό και η συμπερίληψη των Ρωμά είναι απάντηση σε αυτή την ερώτηση μέσω της έκθεσης της κυρίας Γιαρόκα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το περασμένο Οκτώβριο ακριβώ έκανε μια συνεδρία σε υψηλό επίπεδο για να απαντήσει στην ίδια ερώτηση και να δώσει μια απάντηση στην ε, κοινωνικό αποκλεισμό των ε, Ρωμά. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχολείται με το θέμα αυτό από το 1960 και έχει αναπτύξει διάφορα προγράμματα και αρκετή εμπειρογνωμοσύνη. Η συνεδρία υψηλού επίπεδου που, συνεργα... που συνδιοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση εστίασε στις μελλοντικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και συμφώνησε να δουλέψει για κάποια πρακτικά ζητήματα που θα δώσουν ορατά αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα από τα κύρια μέσα είναι, μέτρα είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για, για μεσολαβητές στα σχολεία, στην απασχόληση και στην υγεία. Το πρώτο σχετικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2011 και θα βασιστεί σε προηγούμενη εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε υπάρχον ε, εκπαιδευτικό υλικό, αλλά θα βασίζεται σε νέα ύλη που θα επικυρωθεί από εμπειρογνώμονες μέχρι το τέλος του χρόνου. Κατάρτιση των νομικών θα βασιστεί στα 15 χρόνια ε, εμπειρία του, Ευρωπαϊκού, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για πρόγραμμα το οποίο γίνεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι οργανώσεις των Ρωμά. Επίσης είναι σχεδιασμένο ώστε να επεκτείνει τις συνεχιζόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για δικαστές, εισαγγελείς και αστυνομικούς από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την νομολογία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το δίκαιο για τους ταξιδιώτες αλλά και για τις αρχές κατά των διακρίσεων. Η δήλωση του Στρασβούργου δεν περιορίζεται βέβαια στην κοινωνική διάσταση. Οι πρωτοβουλίες του Στρασβούργου που παρατίθενται στην δήλωση καλούν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την γνώση της ιστορίας των Ρωμά στα σχολεία και να συμπεριλάβουν ε, τους Ρωμά στα ε, σχολική ύλη καθώς και να ενημερώσουν για την ε, κουλτούρα και τον πολιτισμό των Ρωμά, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή πολιτιστικών ε, θεσμών, τοπικών κοινοτήτων, καθώς και καταβλισμών των Ρωμά σε, αυτόν, σε αυτή την προσπάθεια. Ένα άλλο μέτρο που προτείνεται σε αυτή τη δήλωση του Στρασβούργου είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα είναι λειτουργική μέσα στο πρώτο ήμιση του 2011. Αυτό θα βελτιώσει τη δυνατότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης να συλλέγει, να αναλύει, να ανταλλάσσει και να διαδίδει πληροφορίες για πολιτικές και καλές πρακτικές για τους ε, ταξιδιώτες Ρωμά. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συντενή συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, αυτούς δηλαδή που τακτικά συλλέγουν στοιχεία στους τομείς αυτούς. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και η εφαρμογή τους, η δήλωση του Στρασβούργου βασίζεται σε διευρυμένη συνεργασία και συντονισμό ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, σε περιλαμβανωμένο των ενώσεων των Ρώμα. Να προσθέσω στο πλαίσιο αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα τέτοιας ε, συνεργασίας που προηγείται της δήλωσης του Στρασβουργού, δεν είναι αποτέλεσμά της, είναι κάτι το οποίο έγινε παλιότερα, μια παλιότερη πρωτοβουλία και είναι η Διεθνής Task Force για την εκπαίδευση των Ρώμα που πρόσφατα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΣΑ, την UNESCO, τη UNICEF, το Ίδρυμα Εκπαίδευση των Ρωμά και τον Διεθνή Οργανισμό εκπαίδευσης. Βασικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι Ρωμά με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να δελτιωθεί η εφαρμογή του προγράμματος αυτού σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό και διεθνές. Η πρωτοβουλία στο Στρασβούργο καλεί, τα κρατου, καλούν τα κρατημέλη να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τοπικές και εθνικές, περιφερειακές αρχές να εμπλακούν σε πανευρωπαϊκή συνεργασία ανάμεσα σε περιφέρειες και πόλεις με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ε, κοινωνικό και οικονομικό, οικονομική ένταξη των Ρώμα. Ε, με τα χαράς διαπίστωσα ότι το σχέδιο έκθεση της Κομισιόν κάνει παρόμοια έκκληση όταν ζητά από την Επιτροπή να συνεργαστεί με άλλα θεσμικά όργανα, κράτη-μέλη, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διεθνή προγράμματα και ε, οικειό. Τέλος, ενημέρωση θα γίνεται βασιζόμενη στην καλή προηγούμενη εμπειρία της εκστρατείας Ντόστο που έχει γίνει μέχρι στιγμής στα 15 κράτη-μέλη. Είναι μια εκστρατεία κατά των διακρίσεων, κατά τον Ρωμά. Ντόστα θα πει φτάνει. Η αυτή έγινε στη Βουλγαρία και στην Ιταλία και σε διάφορες γαλλικές κοινότητες το 2010 και το 2011 θα επεκταθεί στη Γερμανία, την Ισπανία, στο Κωσυφοπαίδιο και αλλού. Για να διευκολυνθεί η στρατηγική μετατροπή του προγράμματος δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες Ρωμά θα αποτελούν τώρα ένα χωριστό πρόγραμμα που θα αποκαλείται πρόθεση το ρομά κοινωνική ένταξη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο πλαίσιο του προγράμματο δραστηριοτήτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη και θα τοποθετηθεί υπό τον πυλώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση γιατί επιβεβαιώνει ότι τα θέματα που αφορούν το Ρωμά, τους Ρωμά είναι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να διεξασφαλιστεί η οριζόντια προσέγγιση θα βασιστούμε σε οργάνωση ένα πρόγραμμα υπό την ευθύνη του κ. Σάκη Μπρούκ, ενό ε, Ολλανδού νομικού που έχει διοριστεί ειδικό εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για θέματα Ρωμά. Βασικός στόχος για αυτόν τον εσωτερικό διοργα... ε, της εσωτερικής ε, οργάνωσης είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι Ρωμά θα επωφεληθούν πλήρως από την ευρυγνωμοσύνη του οργανισμού και ότι όλα θα γίνουν με συντονισμένο τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, είναι άποψή μας και πιστεύω ότι είναι και άποψη του σχεδίου έκθεσης για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια στρατηγική για την Ευρώπη σημαίνει ευθύνη όλων των κρατών μελών τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά. Δεν πρόκειται για μια ιδεαλιστική στρατηγική, για μια αναφηρημένη έννοια Ευρώπης, αλλά πρόκειται για μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που στόχο έχουν του Ευρωπα... Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι στερούνται των δικαιωμάτων τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, αγαπητέ κύριε. Όλοι μας εκτιμούμε τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μιλήσατε και για την πρωτοβουλία του Στρασβούργου ε, προς όλα τα κράτη-μέλη και τις σχετικές οργανώσεις για να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία με τις εκστρατείες ευαισθητοποίησεως κλπ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για όλες αυτές τις προσπάθειες που ήδη έχετε καταβάλει και βεβαίως ζητούμε τη συνεργασία μαζί σας. Η τελευταία παρέμβαση τώρα θα είναι του κυρίου Ιβανόφ. Καλώς ήρθατε. Από το Περιφερειακό Κέντρο της Μπρατισλάβα του UNDP. Ε, θα σας δώσω μέσα τον λόγο. Μετά από την δική σας παρέμβαση θα ε, διεξαχθεί σύντομη συζήτηση και παρακαλώ Γνωρίστε μας εάν θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι η ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες των Ρώμα είναι θέμα προτεραιότητας. Είναι και θέμα επίσης όπου το κενό, η απόσταση ανάμεσα στις πολιτικές δηλώσεις και υποσχέσεις από τη μια μεριά και ε, την πραγματική πρόοδο ε, επιτόπου, στην πράξη δηλαδή, είναι μεγάλο το κενό αυτό. Χρειάζεται λοιπόν όχι πλέον πολιτικές δηλώσεις, αλλά πράξεις. Και ελπίζω ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω επίσης ότι οι λίγες σκέψεις που θα θέσω υπόψη σας θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί το χάσμα αυτό. Τα περισσότερα από όσα θα πω έχουν ήδη λεχθεί από άλλους σε διάφορες άλλες οργανώσεις ή οργανισμούς, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επαναλάβω ορισμένα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ευθύνη. Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρώμα στην Ευρώπη είναι δύσκολο θέμα. Είναι περίπλοκο και κυρίως λόγω του επίπεδου στο οποίο πρέπει ε, να ε, τοποθετηθεί. Νομίζω ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να σχεδιαστεί με πολύ προσεκτικό τρόπο ώστε να μην προκαλέσει την εντύπωση ότι οι Βρυξέλλες αναλαμβάνουν το θέμα, δηλαδή το παίρνουν από τα χέρια των κρατών μελών για να το φέρουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερο είναι το ζήτημα της ε, γενικότερης αντίληψης ε, για την παρεμβασία αυτή. Ε, ο αποκρισμός των Ρώμα είναι στην πραγματικότητα στέρηση ευκαιριών και εξέλιξης, ανθρώπινης εξέλιξης, που σημαίνει ότι έχει κανείς ελευθερίες και επιλογές, ώστε να ζήσει την ζωή που θεωρεί ότι αξίζει. Στον πυρήνα λοιπόν των προσπαθειών μας θα πρέπει να μπει η δυνατότητα να έχουν οι ε, Ρωμά επιλογές. και όχι από την σκοπιά της εθνικής, εθνοτικής μάλλον ε, ομάδας, ανεξαρτήτως του ποιος αποκλείεται του ποιος είναι φτωχός. Ε, είναι αλήθεια ότι ίσως η πλειοψηφία των Ρώμα είναι φτωχή και αποκλεισμένη. Όχι όμως όλοι. Μιλώντας για τον αποκλεισμό των Ρώμα, αν εμείς με εκείνους, τους Ρώμα, που είναι ήδη ενταγμένοι, έχουν επαγγελματικέ σταδιοδρομίες. ακούμε συχνά ότι οι Ρώμα δεν πρέπει να θεωρούνται σαν μια υποομάδα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι το αντίθετο. Σαν μια μειονεκτική τάξη δηλαδή. Οι λίγες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι σχετικά με την έννοια της ε, συμπερίληψης ή της ένταξης. Ίσως πρέπει να τοποθετηθεί διαφορετικά. Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Ρώμα την συμπερίληψη αυτή και πώς την αντιλαμβάνονται αυτοί που δεν είναι Ρώμα έχω την εντύπωση ότι συχνά οι έννοιες αυτές δεν επικαλύπτονται, δεν είναι ταυτόσιμες. Η διευκρίνηση λοιπόν θα καταστήσει δυνατόν και να τεθούν ερωτήσεις αλλά και να απαντηθούν και κυρίως ποια είναι, ποιο είναι το τίμημα που δέχεται και η μία και η άλλη πλευρά να πληρώσει για την συμπερίληψη των Ρώμα. Εγώ θέτω το ερώτημα διότι η συμπερίληψη, η ενσωμάτωση είναι μια περίπλοκη διάδραση όπου και οι δύο πλευρές κάτι κερδίζουν αλλά και κάτι θυσιάζουν. Είναι μια ε, παράλληλη κίνηση και πολύ συχνά όμως φαίνεται ορισμένοι θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να είναι όμως μονόδρομος κατά τη γνώμη μου. Τέλος, μια τέτοια στρατηγική αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία για να καθοριστούν ποια είναι εκείνα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και ποια πρέπει να αποφευχθούν. Μπορεί να μεταφερθεί πλέον και σε λεπτομερέστερες στρατηγικές. Οι βασικές αρχές της ε, ενσωμάτωσης των Ρώμα αποτελούν σωστή αφετηρία και μπορούν να τις επεξεργαστούμε περισσότερο. Μπορούν να αντιμετωπιστούν ως η βάση για την αξιολόγηση κάθε παρέμβασης για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να οδηγούν σε εξάρτηση, δεν θα πρέπει να αποκλείουν στη βάση εθνοτικής ε, ε ή ε, άλλων τέτοιων χαρακτηριστικών. Οι προτεραιότητες πρέπει να δίνονται, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη σε περιοχές όπου κατοικούν οι Ρώμα. Να δοθεί δυνατότητα της συμβίωσης Ρώμα και μη Ρώμα γιατί αν να βελτιωθούν οι συνθήκες ευημερίας τόπου των τοπικών κοινωνιών είναι το καλύτερο για να μπορέσουν και να ενσωματωθούν και οι Ρώμα σε αυτές. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη της κάθε μελλοντική στρατηγική. Τέλος, η δεκαετία της ε, ένταξης των Ρώμα γνωρίζετε για την πολιτική αυτή πρωτοβουλία. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι κινείται εκ παραλίλου με άλλες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι αυτή η δεκαετία είναι μια μοναδική ευκαιρία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή που προσφέρει για την ανάπτυξη και των μελλοντικών στρατηγικών. Αυτά τα λίγα σχόλια, λίγες σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ως εμπειρογνώμων της UNDP ελπίζω ότι θα μπορέσω να συμβάλλω και περαιτέρω στη συζήτησή σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας κύριε Ιβάνοφ. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στις βασικές αρχές ότι οι Ρωμά είναι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως ε, οι υπόλοιποι πολίτες και είναι σημαντικό το θέμα των ευθυνών, το οποίο συζητήσαμε και χθε. Οι ευθύνε λοιπόν που έχουν τα κράτη-μέλη, την πρωτογενή ευθύνη, α το πούμε έτσι, αλλά και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την ευθύνη καλύτερου συντονισμού και της εδραίωσης μηχανισμών παρακολούθησης της πρόοδου που επιτελείται στα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε σε αυτές τις δύο μέρες της ακρόασης. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ε, που έκαναν παρουσιάσεις και έχουμε λίγο χρόνο, όχι πολύ, για κάποιες ερωτήσεις και σχόλια. Ο κύριος ε, Ιωάννης από τη UNICEF είπε ότι ήθελε να πει κάτι και φυσικά και η, η Λίβια Γιάροκα μπορεί να θέλει να θέσει κάποια ερωτήματα. Η... Παρακαλώ. Και η Κορνέλια Ένστε επίσης μετά. Κάποιος άλλος. Ο Γιώχανες Βέντενικ που ζήτησε το λόγο καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γιώχανες ε, Βέντενικ, είμαι επικεφαλής του γραφείου της ε, UNICEF στο Κωσυφοπαίδιο. Θα ήθελα να διευρύνω λιγάκι τη συζήτηση και στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη και τις χώρες που είναι σε προένταξιακή ακόμα φάση. Έχουμε το θέμα των παιδιών που έφυγαν από τα Βαλκάνια να έρθουν στη Γερμανία. Η UNICEF έκανε μία μελέτη για την ζωή των παιδιών αυτών που είναι παιδιά από το Κόσοβο και Ρώμα στη Γερμανία. Έκανε αυτή τη μελέτη για την ευμάρεια των παιδιών. Η μελέτη κατέδειξε ότι είναι κάπως επισφαλής η αποδοχή αυτών των παιδιών, αλλά είναι καλά ε, ενσωματωμένα αυτά τα παιδιά και ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα Αφού γύρισαν τα παιδιά αυτά στο κοσμοπέδιο, τα δύο τρίτα δεν πήγανε στο σχολείο στη συνέχεια, τα 40% δεν καταγράφηκαν στους, ε, στα δημοτολόγια και οι οικογένειες οι οποίες ε, επανήλθαν από τη Δυτική Ευρώπη ζούσαν σε ακόμα χειρότερες συνθήκες από τις οικογένειες που είχαν μείνει στο Κόσοβο και δεν έφυγαν ποτέ από εκεί. Παρουσιάσαμε αυτή την έκθεση και στη Γερμανική Bundestag και χαίρομαι και για ορισμένε από τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα τώρα. Το κύριο θέμα είναι αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται το καλύτερο συμφέρον του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά το ερώτημα είναι αν έχει νόημα στη συζήτηση που διενεργούμε εδώ, αν έχει νόημα να επαναπατρίσουμε τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία σε καλές συνθήκες και να τα ξανα φέρουμε στο κοσμοπέδιο όπου ουσιαστικά δεν θέλουν να μείνουν, θέλουν απλώ να επιστρέψουν στη Γερμανία. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι δεν ήταν προ το συμφέρον του. Να προσθέσω κάτι. Ξεκινήσαμε, η Κονέλη Ένστε, ξεκίνησε μια γραπτή δήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει ακόμα υπογραφή. Ελπίζουμε να συλλέξουμε και περισσότερες υπογραφές για το θέμα αυτό γιατί αυτό είναι μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση. Η Λίβια, αν θέλει να λάβει το λόγο τώρα, χωρίς μικρόφωνο η Λίβια. Σε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, ευχαρίστω. Η Κορνέλια τότε. Και μετά η Μπίργκετ. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Χθε και σήμερα με απασχολεί το ίδιο ερώτημα, που μου φαίνεται και ερώτημα κλειδί και κάπως ξεπήδησε και μέσα από τις παρεμβάσεις όσο μπόρεσα να τις παρακολουθήσω σήμερα. Τι μπορεί να γίνει, πραγματικά δηλαδή, στην πράξη, χωρίς λόγια, ώστε η Ρώμα από την αρχή, από την αρχή να συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή αλλαγών. Από την αρχή, αυτό τονίζω. Δηλαδή ανησυχώ ότι καθόμαστε εδώ, εκφράζουμε σκέψεις πολλές για τους Ρώμα, μειώντας Ρώμα ίδιοι. Και ίσως και χωρίς να το θέλουμε, παίρνουμε μια στάση πατερναλιστική. Επαναλαμβάνω, χωρίς να το θέλουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ποιες είναι οι δομές που θα έπρεπε να επιλέξουμε στις χώρες μέλη, αυτό είναι το ερώτημα που θα ήθελα να κάνω, που θα ήταν και σκόπιμες και που από μιας αρχής θα επέτρεπαν ε, την συμπερίληψη, την συμμετοχή των οργανώσεων Ρώμα. Ποιες δυνατότητες δηλαδή μπορούν να δημιουργηθούν. Να μπορούν να μας πούν οι Ρώμα αυτά που πάτε να κάνετε μπορεί να είναι από καλή θέληση αλλά είναι λάθος και θα έπρεπε να κάνετε το ΑΒΓ. Είμαι πεπισμένη ότι όλα όσα μετά θα δημιουργήσουμε ή θα κάνουμε για τους Ρώμα, αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα είναι αυτά τα πράγματα που θα θέλαν οι ίδιοι. Το ίδιο, η ε, αντίστοιχα, θα ήταν και για άλλες ομάδες, για τις γυναίκες για παράδειγμα. Γι' αυτό το ερώτημα που με απασχολεί είναι ποιες δομές θα πρέπει να δημιουργηθούν στην πράξη μέθοδοι, μηχανισμοί στα κράτη-μέλη, ώστε οι ε, Ρώμα να συνδιαμορφώσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι για μένα το πιο κεντρικό ερώτημα. Όλα τα άλλα νομίζω τα συζητήσαμε λίγο πολύ και χθε. Η Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ Κονέλια, πράγματι πρόκειται για το πιο θεμελιώδες ερώτημα και η ακρόαση αυτή είναι μέρος του διαλόγου αυτού. Μπέγκης πάλι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω πρώτα τις ε, δηλώσεις ε, του Επιτρόπου Άγγε. Όταν μιλούμε για ενσωμάτωση ή ένταξη, πρέπει να είναι συνολική προσέγγιση, δηλαδή σε πολλούς τομείς. Από την εκπαίδευση μέχρι τη στέγη, μέχρι το επάγγελμα, την επαγγελματική δραστηριότητα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ταυτόχρονα βέβαια με ποια βαρύτητα θα αντιμετωπιστούν οι διάφοροι τομείς. Αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το περιφερειακό ή τοπικό πλαίσιο, ώστε η συνεργασία όχι μόνο με τις χώρες μέλη, αλλά και με τους τοπικούς φορείς είναι πάρα πολύ σημαντική και ιδίω, και όταν μιλούμε για το πώς θα συνδιαμορφωθούν διάφορα project μαζί με τους ενδιαφερόμενους. Εμένα μου φαίνεται σημαντικό το ερώτημα αυτής της συνεργασίας με, με τους τοπικούς φορείς. Ποιες δυνατότητες έχουμε όμως να ελέγξουμε, να ενθαρρύνουμε και όλα στους τοπικούς φορείς, ώστε πραγματικά να εφαρμοστούν αυτά τα ε, σχέδια. Διότι όσο θαυμάσια και να είναι αυτά που θα συζητήσουμε και θα εκπονήσουμε εδώ, δεν πρόκειται να ωφελήσουν τίποτε εάν δεν εφαρμοστούν τελικά επιτόπου. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Αν μπορέσουμε να επιτύχουμε ιδίω για την ενσωμάτωση των Ρώμα ως μεγάλης, πολύ μεγάλη μειονότητα να προχωρήσουμε και κάτι τέτοιο θα είναι μεγάλη πρόοδος και για τους Ρώμα, αλλά θα ήταν σημαντικό, εφόσον είναι επιτυχές το διάβημα αυτό, να επαναληφθεί και για άλλες μειονεκτικές πληθυσμιακές ομάδες γιατί νομίζω ότι η βελτίωση χρειάζεται σε πάρα πολλούς τομείς. Σας ευχαριστώ και εσάς ιδιαίτερα. Μένει η Μιράντα Μολασφάντα από το φόρουμ Ρωμά της Φιλανδίας. Α, έχει, έχει αποχωρήσει. Α, είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαστε στη βάση της συζήτησης που μιλάμε για την ευρωπαϊκή στρατηγική των ε, Ρωμά ή για την ευρωπαϊκή στρατηγική πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές, όπως και να το περιγράψετε. Αυτό μας ενδιαφέρει δεν είναι το όνομα, αλλά το περιεχόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σικλούνα ένα ερώτημα. Όταν μίλησατε για τη δήλωση του Στρασβούργου και την εκπαίδευση των ομομαθών και των διαμεσολαβητών για τους Ρωμά, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν, ποιοι είναι η ομάδα στόχων που θέλετε να αντιμετωπίσετε για αυτές τις λειτουργίες. Είναι Ρωμά ή δεν είναι Ρωμά, είναι και, και, και Ρωμά και μη Ρωμά. Και μέσα σε αυτή τη δομή που θέλετε να δημιουργήσετε, ποια θα είναι η εντολή αυτών των ανθρώπων, ποιος θα είναι ο ρόλος τους, ποιος θα τους δώσει εντολή, με ποιο τρόπο θα διεισδύσουν στις κοινότητες σε εθνικό επίπεδο το Ρωμά και θα παίξουν κάποιο ρόλο διαμεσολαβητικό μεταξύ των δημοσίων αρχών και των κοινοτήτων το Ρωμά για να μπορούν οι κοινότητες αυτές να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στα θέματα που τους εμπλέκουν. Ελέγχθη από κάποιον ο κ. Ιβάνοφ, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ενσωμάτωση των Ρωμά στην Ευρώπη πρέπει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση για την αύξηση της ε, συνειδητοποίησης τόσο το Ρωμά όσο και των μη Ρωμά. Και αυτό ανέφερε και ο Επίτροπος Αντόρ, τόνισε ότι ένας από τους λόγους της, ε, του αποκλεισμού το Ρωμά από την πολιτισμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα είναι ότι για χίλια χρόνια και παραπάνω η Ευρώπη έχει θέσει στο περιθώριο τους Ρωμά και έχει παραγνωρίσει την παρουσία του εδώ. Εγώ ήμουνα δασκάλα. 18 χρόνια ήμουνα δασκάλα στο σχολείο. Έχουμε ίσως ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στην Φιλανδία και σε, πολλές, σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς και συγκρίσεις έχουμε έρθει πρώτοι, αλλά ακόμα και στη Φιλανδία. Για να μην μιλήσω για άλλες εκπαιδευτικές δομές στην Ευρώπη, δεν υπάρχει μία τέτοια κατάσταση που να εξασφαλίζει την αναγνώριση των Ρωμά στα εκπαιδευτικά υλικά, στο σχολικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για τους Ρωμά και αν δεν ενσωματωθεί στα σχολικά προγράμματα, οτιδήποτε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε με σχέδια στρατηγικής, με στρατηγικές, όλα αυτά δεν πρόκειται να βοηθήσουν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, γιατί τελικά είναι το θέμα της αντίληψη το οποίο έχει σημασία και η αντίληψη αυτή, η αρνητική για τους τσιγκάνους που βρίσκεται στην Ευρώπη, αυτή πρέπει να καταπολεμηθεί. Επομένως, η αύξηση της συνειδητοποίησης είναι ένα από τα κύρια θέματα, αλλά δεν είναι από μόνη της επαρκής, είναι απλώς ένα σημείο εκκίνησης. Θα πρέπει να υπάρξει μια δομή η οποία θα διατρέχει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, το να υπάρξει αναγνώριση των Ρωμά ως μιας ιστορικής μειονότητας της χώρας μας. Αν δεν γίνει αυτό από επίπεδο παιδικού σταθμού μέχρι επίπεδο πανεπιστημίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε σε 20 χρόνια ίσως να έχει αλλάξει η κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη. Γιατί όλα εξαρτώνται από την αντίληψη που έχουν αυτοί που είναι σε θέσεις Λήψη αποφάσεων και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευτεί να βλέπουν του Ρωμά σαν ισότιμους Ευρωπαίου πολίτε δεν πρόκειται να κάνουν τι απαραίτητε αλλαγέ ακόμα και να ακολουθήσουν σωστέ στρατηγικές. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στα θέματα αυτά, γιατί δεν πρόκειται μονάχα για τις λήπτες αποφάσεων. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτές τις συμβολές και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους ομιλητές αν θέλουν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά που ελέγχθηκαν. Κύριε Άντορ. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να δώσω μια σύντομη απάντηση γιατί ακόμα και σε μια σύντομη απάντηση θα πρέπει να αντιμετωπίσω πολύπλοκα θέματα. Να ξεκινήσω από το τέλος. Θέσατε το θέμα της συνειδητοποίησης και της αντίληψης που έχει για τους Ρωμά η πλειοψηφία. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόναχα για τις χώρες που είναι τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Ρωμά, αλλά και εν γέννη. Ίσως γνωρίζετε τον Γκούναρ Μίρνταλ, το γνωστό Σουηδό οικονομολόγο. Στην δεκαετία του 1940 αντιμετώπισε το πρόβλημα της μειονότητας των μαύρων στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είπε ότι λίγο μετά από την ε, εκκίνηση της έρευνάς του, ε, είπε ότι δεν νομίζω ότι η Αμερική έχει πρόβλημα με τους μαύρους, έχει πρόβλημα με τους λευκούς. Έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση εδώ. Και συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό η συζήτηση δεν πρέπει να εστιάζεται, η συζήτηση για τους Ρώμα δεν πρέπει να εστιάζεται μονάχα Ρώμα. Χρειαζόμαστε μια γενικότερη πολιτική κατά των διακρίσεων, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα, γιατί υπάρχουν και ε, Ρώμα που έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση, έχουν υψηλό εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά ακόμα και αυτοί αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα παιδείας, τα άτομα αυτά δεν επιλέγονται για θέσεις υψηλής ευθύνης λόγω αυτή τη διάκριση που ασκείται εναντίον του. Αυτή είναι λοιπόν μια διάσταση, μια άλλη διάσταση <coughs> την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στην οποία εστιάσαμε ιδιαίτερα είναι το θέμα τη εξάρτηση τη ένδυα. Γιατί η ένδυα το Ρωμά είναι τέσσερι φορέ πιο διαδεδομένη από ό,τι στο γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό. Αυτό είναι σημαντικό, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα των διακρίσεων, της περιθωρικοποίησης, της έλλειψης παιδείας, της έλλειψης πρόσβασης στη στέγαση, της έλλειψης ευκαιριών για τους Ρωμά. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να σπάσει αυτόν τον κύκλο, Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η προσπάθεια να συνενώσουμε τις πολιτικές μας, να φέρουμε από κοινού όλους τους εμπλεκόμενους και να ενισχύσουμε και τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την κυρία Ένστε, ότι είναι κέριου χαρακτήρα η συμμετοχή. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα μόνο με χρηματοδότηση και με την παροχή ευκαιριών. Όταν πήγα στο Βουκουρέστι, εγώ συναντήθηκα με τους ηγέτες ομάδων Ρώμα που ήταν ενεργοί, προσπαθήσαν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου, πολλές φορές απέτυχαν, δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στα αυτά κονδύλια. Επίσης συναντήθηκα με τους Ούγγρους ηγέτες των Ρωμά και συνεχίζω αυτές τις προσπάθειες γιατί η ανάδραση από, τη, από τους Ρωμά είναι πολύ σημαντική για μας για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μελλοντικά προγράμματα και το μελλοντικό κανονισμό των διαδοτικών πόρων. Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που προωθούν την απλοποίηση για το κοινωνικό ταμείο. Έχουμε πολύ περιθώριο ακόμα για απλοποίηση στα θέματα αυτά και τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εύκολα προσβάσιμα για όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση περιθωρικοποίησης και έλλειψη εμπειρίας με τη διαδικασία χρησιμοποίησης αυτών των πόρων. Γι' αυτό εμεί θα πρέπει να προσαρμόσουμε το σύστημα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να την χάνει καλύτερες χρήσεις και συμφωνώ με τον κύριο Ιβάνοφ για τη σημασία του να θεσπίσουμε προγράμματα που δεν έχουν εθνοτικά αποκλειστική προσέγγιση γιατί πρέπει να βοηθήσουμε την ε, ανάπτυξη των μικροπεριοχών στις οποίες ζουν οι Ρώμα σε μεγάλους αριθμούς και συγχρόνως την εσωμάτωσή τους στο γύρο κορμό της κοινωνίας. Και αυτό μας φέρνει στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι σε πολλές από τις περιοχές ή μικροπεριοχές όπου διαβιβούν σε, σε μεγάλο πληθυσμό οι Ρωμά στην Ουγγαρία, Ρωμανία, Βουλγαρία και Σλοβακία, αν δεν προωθήσουμε την ε, τοπική οικονομία και τον μη κερδοσκοπικό τομέα, τους συνεταιρισμού και όλες αυτές τις ε, δυνητικά επιδοτούμενες μορφές απασχόλησης, δεν μπορεί να υπάρξει η απαραίτητη τομή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε, να σκεφτούμε περισσότερο και με τους άλλους αρμόδιους ε, επιτρόπους, αλλά προσπαθούμε και με, την, ε, με τον Νταλή, με τον Μπαρνιέ, με άλλους επιτρόπους, προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Είναι μια σημαντική κατεύθυνση λοιπόν αυτή για μας. Και εν κατακλείδη θέλω να πω ότι από τη στιγμή που θα μπορούμε να αποκομίσουμε μια σαφή εικόνα από τα συμπεράσματα της ε, Task Force, της Δυναμής Κρούσης, ίσως θα είναι σκόπιμο να συναντηθούμε και πάλι και να σας ενημερώσω για τα επόμενα βήματα που προετοιμάζουμε για το πλαίσιο εθνικών στρατηγικών συμπερίληψης των Ρωμά. Γιατί μιλάμε για ένα πλαίσιο, νομίζω το ανέφερε πολύ σαφώς ο κύριος Ιβάνοφ, γιατί η θεμελιώδης ευθύνη πρέπει να παραμείνει στα κράτη-μέλη, γιατί έχουμε να κάνουμε για τους πολίτες των κρατών αυτών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο, ένα ρόλο συντονισμού, με την μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών, των καλύτερων μάλλον πρακτικών, γιατί βελτίωση των πρακτικών είναι κάτι πολύ δύσκολο να το πούμε. Υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές. Παρ' όλα αυτά δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Νομίζω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξαν κάποια θετικά στοιχεία, κάποια πρόοδος η οποία επετέφθη, αλλά είναι καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα και να αυξήσουμε την ταχύτητα των προσπαθειών μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, like... <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπή. Κύριε Σικλούνα, εσείς, αν θέλετε, απαντήστε σε ορισμένες από τις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τους διαμεσολαβητές, δεν πρόκειται για κανένα νέο είδος. Υπάρχουν εδώ και χρόνια οι μεσολαβητές αυτοί. Και στη Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι συνήθις πρακτική. Στη Μολδαβία, επίσης, εισήχθη ο θεσμός, καθώς και σε άλλες χώρες. Άρα, δεν είναι απολύτως νέο <clears throat> το στοιχείο αυτό. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η συνάντηση υψηλού επίπεδου ήταν να αυξήσει την πρακτική και ίσως μάλιστα να αλλάξει λίγο και το νόημα. Διότι μέχρι τώρα ο διαμεσολαβητής σε ορισμένε από τις χώρες ήταν περισσότερο ένα πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως διαιτητής για την επίλυση διαφορών ε, και κυρίως με τα σχολεία, γιατί συνήθως πρόκειται για διαμεσολάβηση ε, στα σχολεία. αυτό, που προσπαθεί να κάνει η διακήρυξη του Στρασβούργου είναι να ε, ενισχύσει και να αυξήσει τον ρόλο των διαμεσολαβητών και να τους προσφέρει και κάποια υποστήριξη. Ο διαμεσολαβητής δεν θα είναι κάποιος πλέον ο οποίος μόνο συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών, αλλά κάποιος που αποτελεί την γέφυρα μεταξύ του σχολείου ή της ε, αρχής δημόσιας υγείας, ε, εάν πρόκειται για θέμα υγείας, και να είναι, όπως είπα, η γέφυρα να παρέχει πληροφορίες και σε σχέση με το σχολείο να υποστηρίξει και τα παιδιά όταν τελειώσουν το σχολείο. Αυτό νομίζω είναι κάτι που γίνεται νομίζω στην Δημοκρατία της Μακεδονίας όπου έχουν κοινοτικά κέντρα όπου οι διαμεσολαβητές ε, δεν είναι μονάχα υπεύθυνοι για να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο αλλά και για να βοηθήσουν τα παιδιά όταν τελειώνουν το σχολείο ή στη διάρκεια των σχολικών ωρών για να κάνουν κάποια δουλειά που αλλιώς δεν θα μπορέσουν να κάνουν είτε διότι κανείς δεν υπάρχει για να τα βοηθήσει γιατί δεν έχουν κάπου να κάνουν τα μαθήματά τους, δεν έχουν χώρο. Ε, αυτά κάπως είναι τα καθήκοντα των διαμεσολαβητών. Θα ήθελαν να τα επεκτείνουν και σε πολλά άλλα πράγματα και στις δημόσιες υπηρεσίες ώστε ο διαμεσολαβητής να μην είναι μονάχα κάποιος που βοηθάει λίγο είτε στην εκπαίδευση είτε στην υγεία αλλά και σε άλλους τομείς σε τρόπο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν βοήθεια, για παράδειγμα, σε πολλά γραφειοκρατικά ε, θέματα. Σε ό,τι αφορά το ποια θα πρέπει να είναι τα πρόσωπα αυτά των διαμεσολαβητών, εμείς επιμείναμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας και της παιδείας, Επιμείναμε λοιπόν ότι οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι Ρώμα και όχι κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, ίσως αυτό μπορεί να συζητηθεί. Αλλά για τα δύο αυτά θέματα, παιδεία, υγεία, τονίσαμε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να είναι Ρώμα, όπως είπα. Αυτό βέβαια βρίσκεται ακόμα στη φάση της προπαρασκευής. Έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, αλλά το πώς θα λειτουργήσει τελικά δεν το γνωρίζουμε ακόμα είναι και το θέμα πόσοι θα εκπαιδευτούν, γιατί δεν έχει νόημα να εκπαιδεύσετε εκατοντάδες διαμεσολαβητών, εάν δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δουλειά ως διαμεσολαβητές. Δεν είναι απλοί εθελοντές, είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να ασκήσουν μια επαγγελματική δραστηριότητα και άρα θα πρέπει να αμείβονται. Θα πρέπει επίσης να αποφασιστεί ποιος τους πληρώνει και πόσοι εξ αυτών όντω είναι αναγκαίοι. Πάντως συζητούνται τα θέματα αυτά. Ο Γενικό Γραμματέα επιθυμεί να προχωρήσει ταχύτατα, γιατί πιστεύει, όπως και οι περισσότεροι νομίζω από εμά εδώ, ότι πολλή χρόνος έχει περάσει και πολλή χρόνος έχει χαθεί και κάτι πρέπει να γίνει το δυνατόν συντομότερο. Αλλά βέβαια όλοι γνωρίζετε επίσης ότι συχνά όταν κανείς βιάζεται πολύ μπορεί να κάνει και πολλά λάθη. Και ελπίζω να το αποφύγουμε αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιβανόφ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ο χρόνος τρέχει. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα αν αφορά την κάπως πατερναλιστική προσέγγιση. Πολλές συχνά όντως πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Κάνουμε κάτι για τους Ρώμα και από πλευράς των Ρώμα χωρίς τους ίδιους. Και αν και επαναλαμβάνουμε διαρκώς ότι τίποτα δεν πρέπει να γίνεται για τους Ρώμα χωρίς τους ίδιους, τελικά δεν ε, απομακρυνόμαστε από αυτή την πατερναλιστική συνήθεια. Νομίζω πως το κλειδί είναι να δούμε το θέμα μέσω της προοπτικής των ευκαιριών. Θα πρέπει δηλαδή να δοθούν ίσες ευκαιρίες ώστε να ε, μπορέσουν να ασκήσουν το πλήρες τους δυναμικό και τις ελευθερίες τους. Γιατί διαφορετικά ε, διαρκώς ε, πέφτουμε στην ίδια παγίδα. Μιλάμε για τις καλές πρακτικές, αλλά κάποιες φορές θα πρέπει να δούμε τις κακές πρακτικές. Τι δεν λειτουργεί δηλαδή και τι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι γιατί τίνουμε να αναφέρουμε όλη την επιτυχία, γιατί διαφορετικά γιατί βρισκόμαστε εδώ. Αλλά ίσως κάποιες φορές θα πρέπει να βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Πιστέψτε με ότι θα έχουμε πολλά σημαντικά διδάγματα να αποκομίσουμε από μια τέτοια προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη μας ε, συζήτηση και να ζητήσω από τους ομιλητές την κυρία Ιζαμπέλ Μιχελάς, την κυρία Ανδριάννη Παπαδοπούλου, Πρώτη μας ομιλήτρια είναι η κυρία Ιζαμπέλ με χαλάσε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ αντιπροσωπεύω τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που βρίσκεται στην ε, Ουγγαρία. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διαδικασία της στρατηγικής Ρωμά για την ε, κοινωνική ένταξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα χτες θα ακούσατε από πολλούς συναδέλφους και κυρίως από την κυρία Λίβε Γιάροκα, Άρα κάποια πράγματα θα τα επαναλάβω, αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η θέση μας όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Τον, ε, στα τέλη του Ιανουαρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ψήφισε ένα ψήφισμα για ε, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά, σημειώνοντας ότι οι Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουν από ρατσιστικές διακρίσεις, πολλές φορές υπόκειται σε αυστηρή διαρθρωτική διακρίσεις, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και πολλαπλές διακρίσεις επί τη βάση του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ισότητα των Ρωμά έχουν αποτύχει να δώσουν οποιοδήποτε σημαντική βελτίωση στι κοινότητε των Ρωμά αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμα αντιμετωπίζουν οι Ρωμά διακρίσεις θεσμικέ, υψηλά επίπεδα φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώ και διακρίσει στη στέγαση, στην παιδεία και στην υγειονομική περίθελψη. Ε, γίνονται επιθέσεις ε, βίες, ε, ρατσιστικές, καθώς και αστυνομικές επιδρομές. Όλα αυτά τα βλέπουμε στους τίτλους των εφημερίδων. Η αδυναμία να καταδικάσουμε του είδους αυτό το λόγο κατά τον Ρωμά ε, τελικά παραβιάζει το κράτο δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανάγκη για ύπαρξη Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρωμά έχει διαπιστωθεί από πολλές ΜΚΟ, διεθνεί οργανισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ θέλω πάλι να ευχαριστήσω την κυρία Λίβα, Λίβια Γιάροκα για την ε, σπουδαία πρωτοβουλία που ανέλαβε για την στατηγική για το Ρωμά και την κοινωνική, και τους ένταξη, που βρίσκω ότι είναι εξαιρετική πρωτοβουλία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί φαίνεται να μην έχουν μια συμπαγή στάση και να δίνουν λαβή για διάφορε ερμηνείε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει αυτό το ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και την ε, Κοινωνική Ένταξη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για εθνικέ ε, στρατηγικέ για του Ρωμά. Εμεί πιστεύουμε ότι άσχετα από το τίτλο, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ω αποτέλεσμα μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα μεγιστοποιεί τους πόρους για την ένταξη των Ρωμά, που θα θεσπίζει κάποιες γενικές απαιτήσεις για την προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρωμά και που θα απαιτήσουν από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν συγκεκριμένες ε, ε, όρια για την, ε, για, για την ένταξη. Γι' αυτό μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι συνεπής, συμπληρωματική, καθώς και να ε, αποτελεί ένα μέσο συντονισμού ώστε να υπάρχει αποτελεσματική στόχευση των Ρωμά. Αν θέλουμε λοιπόν η Κομισιόν δηλαδή να αποτελεί το σημείο συντονισμού των προσπαθειών και να καθοδηγεί τα κράτη-μέλη στις εθνικές τους στρατηγικές. Γι' αυτό το σκοπό μια μόνιμη task force θα πρέπει να δημιουργηθεί γιατί για την ώρα είναι προσωρινή και θα πρέπει να έχει το ρόλο συντονιστικό για την στρατηγική να θεσπίζει, ε, να κάνει μάλλον συγκρίσεις και να παρακολουθεί την πρόοδο καθώς και να αναφέρει την πρόοδο της στρατηγικής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική συμμετοχή ε, ε, υψηλά ισταμένων υπαλλήλων από τα κράτη-μέλη, από τους θεσμούς, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Προεδρία κάθε φορά, ώστε να γίνεται ανταλλαγή των καλών πρακτικών και της εμπειρογνωμοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τις υποψήφιες χώρες, και νομίζω ο συνάδελφος από το Κοσυχοπαίδιο τόνισε τη, τη σημασία της ε, συμπερίληψης αυτή τη διαδικασία των χωρών ε, υποένταξη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο συντονισμός με τις υπάρχουσες <coughs> διακυβερνητικές πρωτοβουλίες, ε, την ΟΑΣΕ, την ε, δεκαετία για την ε, ένταξη των Ρώμα, τις στρατηγικές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η στρατηγική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σαφείς στόχους, δράσεις, ε, κριτήρια αξιολόγησης, παρακολούθησης και δείκτες και θα πρέπει να διευκολύνει τους Ρωμά να ιδιοποιηθούν τη βελτίωση της δικής τους κατάστασης και να κυριστούν τους μηχανισμούς που τους απομακρύνουν από την ισότιμη μεταχείριση. Η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στην υποχρέωση των κρατών μελών υπό το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτσι ώστε να δώσουν το πλαίσιο για την ε, κατάργηση των, του αποκλεισμού. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στη στέγαση. Θα πρέπει να έχει στόχο επίσης ε, την ε, καταπολέμηση της ε, καχυποψίας ε, απέναντι στους γύφτους, του θα πρέπει να μπορούν οι Ρωμά να κάνουν συμβάσεις, να προβαίνουν μάλλον σε συμβάσεις, να έχουν ίση και ίδια παιδεία και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα συμβάλλουν στην ε, διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, και η Ένωση να μπορεί να συνδέσει άμεσα τη χρηματοδότηση με συγκεκριμένες δράσεις. Ε, η κοινωνική ένταξη των Ρωμά θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στις ε, πολιτικές της Ένωσης αλλά και στην προγραμματική περίοδο 2014 με 2020. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν μηχανισμοί και διαδικασίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνική ένταξη, της απασχόλησης, τη ισότητα των φύλων, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που επιδιώκουν αυτού τους πολιτικούς στόχους. Να θεσπίσει επίπεδα και δείκτες για να δίνεται η απαραίτητη στήριξη στην έρευνα και στην ε, αξιολόγηση των προγραμμάτων. Η στρατηγική θα πρέπει να απαιτεί μη ομαδοποιημένη συλλογή στοιχείων σε όλους τους τομείς ώστε να μπορεί να γίνει η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. Πολλά κράτη-μέλη, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήδη συλλέγουν ε, στατιστικά στοιχεία υπό διάφορα κυβερνητικά μέτρα, αλλά δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για στόχους επεξεργασίας στοχευμένων πολιτικών προγραμμάτων για συγκεκριμένα προβλήματα. Και θα σας δώσω ένα, ένα παράδειγμα. Σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε σε διάφορες χώρες, διαπιστώσαμε ότι για παράδειγμα στη Ρουμανία η διοίκηση για την υγειονομική περίθεψη διατηρούσε στοιχεία για τα παιδιά και την εθνικότητα των παιδιών, αλλά δυστυχώς αυτά τα στοιχεία ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο. Πιστεύουμε πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απαιτείται να φτιάχνουν ένα πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων παιδείας και επασχόλησης, ας πούμε, για μέχρι το 2020 και αυτό είναι το επίπεδο συμμετοχής αν θέλετε που θα θέλαμε να υπάρχει. Τα κράτη-μέλη δηλαδή να συλλέγουν στις στατιστικά στοιχεία για την ε, παρακολούθηση του σχολείου, για τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, τον αριθμό παιδιών που φοιτούν σε κανονικά σχολεία ή σε χωριστά σχολεία και ούτω καθεξής. Να τελειώσω λέγοντας ότι η στρατηγική θα πρέπει να εξασφαλίσει την ενίσχυση των Ρωμά ως αναγνωρισμένους ε, εταίρους στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών στατηγικών ε, ένταξης των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει θετικά προγράμματα δράσης που προωθούνται από τα ε, ευρωπαϊκά όργανα, τις διάφορους οργανισμούς και συγκεκριμένα κονδύλια για τις ΜΚΟ των Ρωμά, ώστε να παρακολουθούν αυτές τις δραστηριότητε και τα προγράμματα. Στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχει αυτό που λέγεται τεχνική βοήθεια στη δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορεί να εκπονήσει και να εφαρμόσει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διευθυντικά ε, ταμεία. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση που να δίνει προτεραιότητα ή που να δίνει τεχνική βοήθεια στις ΜΚΟ ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση καταρχήν σε ευρωπαϊκά κονδύλια και δεύτερον αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να διευκολύνει τις ΜΚΟ να κάνουν την παρακολούθηση για την εφαρμογή, την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλέσκου, Μιχαλάτσες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συλλογή των απαιτήσεων και των προσδοκιών από τη στρατηγική των Ρωμά. Αυτό το οποίο δεν αναφέρεται πολύ συχνά είναι η συλλογή δεδομένων. Αυτά είναι ένα από τα κέρια θέματα να υπάρξει μια συλλογή δεδομένων η οποία όμως να καλύπτει τις προϋποθέσεις της οδηγίας για την προστασία δεδομένων. Συμφωνώ μαζί σας όμως ότι το να έχουμε πολιτικές οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία θα πρέπει να προωθήσουμε καλύτερα την συλλογή εμπεριστατωμένων στοιχείων. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή που αναφέρατε. Προχωρούμε και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ανδριανή Παπαδοπούλου, η οποία εκπροσωπεί το γραφείο του Έλληνα Διαμεσολαβητή, να μας δώσει τώρα την παρουσίασή της. Έχει το, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Έχοντας παρακολουθήσει τη χθεσινή συζήτηση και έχοντας δει τις απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν χθε, είμαι πεπισμένη ότι μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπερίληψη των Ρωμά θα, έπρεπε, θα έδινε κάποιες κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη και αν είναι δεσμευτική η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά στην κατάσταση των Ρωμά σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Έλληνας διαμεσολαβητής έχει αντιμετωπίσει περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν ε, Ρωμά ήδη από την αρχή της ύπαρξης του γραφείου του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής πήρε το χαρακτήρα ενός φορέα ισότητας από το 2005 και έκτοτε η αρχή του διαμεσολαβητή έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει πιο συστηματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά στην Ελλάδα και να προτείνει προς το κράτος ενέργειες οι οποίες θα προωθήσουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία. Εξετάσαμε μεμονωμένες περιπτώσεις, κάναμε επιτόπιες έρευνες και έχουμε διατυπώσει, έχουμε εκπονήσει και ειδικέ ε, εκθέσεις που περιλαμβάνουν τις προτάσεις μας και φυσικά έχουμε και μία ετήσια έκθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βάσει τη εμπειρία μα, λοιπόν, μπορώ να κάνω τι εξή παρατηρήσει. Καταρχήν, Παρά το γεγονός ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμερίζονται τις ίδιες αρχές για την ίση μεταχείριση των ε, ευάλωτων ομάδων όπως η Ρωμά και γνωρίζουν ποιες είναι οι επιτυχείς πρακτικές για την κοινωνική του ενσωμάτωση, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πραγματική στην πράξη ενσωμάτωση των Ρωμά. Ίσως οι πραγματικές συνθήκες, όχι μόνο οικονομικές αλλά και ιστορικές, πολιτιστικέ και πολιτικές, οδήγησαν σε διαφορετικό επίπεδο βιωτικό και διάφορα ε, στάδια συμπερίληψης των Ρωμά στη, σε κάθε χώρα. Στο Βέλιο Παγκοσχάρη πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καταβλισμοί για τους Ρωμά όπως υπάρχουν στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπερίληψη των Ρωμά πρέπει να είναι αρκετά ευρεία για να επιτρέψει να υπάρξει ανάπτυξη από διαφορετικά αρχικά επίπεδα αλλά συγχρόνως πρέπει να είναι αρκετά αυστηρή για να, επιτρέψει, να, να μην επιτρέψει να υπάρξει αδράνεια από τα κράτη-μέλη και διατήρηση του status quo. Στη χώρα μου, ήδη από τη δεκαετία του 1970 και μετά, υπήρξαν πραγματικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Ρωμά. Είναι όμως πλοκό αυτό το θέμα και μαζί με την έλλειψη μόνιμης προσπάθειας και προσοχής για το θέμα αυτό για την ανάπτυξη των καταλήλων πολιτικών μαζί με την ε, έλλειψη απαραίτητης και ανάλογης σχεδίασης και παροχής πόρων οδήγησε σε επιτυχία που ήταν σπασμωδική και αποσπασματική και μονάχα. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά τη στέγαση του Ρωμά Στην Ελλάδα η κατάσταση τον Ρωμά δεν μπορεί να θεωρηθεί ομοιογενής. Υπάρχουν Ρωμά που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην ελληνική κοινωνία και Ρωμά που ζουν σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού κοινωνικού. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι οι Έλληνες Ρωμά έχουν πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο από τους μετανάστες Ρωμά που έχουν φτάσει στη χώρα μας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Οι απαράδεκτες καταστάσεις όμως στις οποίες ζουν πολλοί Ρωμά στην Ελλάδα μαζί με τις ε, δραστηριότητες της ανεπαρκής που έχουν για να επιβιώσουν έχουν οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες για όλες τις κοινωνίες που ζουν σε καταβλισμούς, κοινότητες στους καταβλισμούς. Επομένως, δεν πρέπει η κυβέρνηση να διαφοροποιεί μεταξύ των Ρωμά επί τη βάση της υπηκότητος αυτών των ατόμων. Αυτό υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι υπάρχει και ε, επιμειξία μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων κινητήτων, δηλαδή των Ιθαγενών Ρωμά και των μεταναστών Ρωμά και επίσης στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά, άτομα τα οποία δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποιος είναι Έλληνας πολίτης και ποιος δεν είναι όταν έχετε ιδίως μεγάλες οικογένειες. Του του οι κύριε πολιτικέ οι οποίε εφαρμόστηκαν τι τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη τα προγράμματα στέγασης, τα προγράμματα εκπαίδευση, οι επιδοτήσει για επιχειρήσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα των Ρωμά, κατευθυνόντουσαν μονάχα προς τους Έλληνες Ρωμά. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι ανεξάρτητα από το βαθμό τη νομική ευθύνη που έχουν τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και του ηθαγενούς πληθυσμού των Ρώμα και των μεταναστών. Φυσικά υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο αυτών βασικών ομάδων <clears throat> στους τέσσερις κύριους τομείς της κοινωνικής ζωής, δηλαδή στη στέγαση, στην παιδεία, στην απασχόληση και στις κοινωνικές παροχές. Για τη στέγαση. <clears throat> Οι Έλληνες Ρώμα που ζουν νομίμως σε μεγάλες πόλεις όπως η Λάρισα δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Τα προβλήματά τους είναι κυρίως να βρουν χώρο για την επέκταση των κοινοτήτων τους. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η αδράνεια, η αρνητική αντιμετώπιση των τοπικών αρχών είναι ένας έμεσος τρόπος διάκρισης σε βάρος τους. Εγώ επισκέφτηκα πρόσφατα τον προηγούμενο μήνα μια κοινότητα στη Βόρεια Ελλάδα όπου δόθηκαν στεγαστικά δάνεια στα μέλη της ε, κοινότητας του Ρωμά. Ήταν πολύ επιτυχή αυτά τα συστήματα σε ορισμένες περιοχές, αλλά όχι σε άλλες. Στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή ερευνήσαμε τα παράπονα ατόμων οι οποίοι είχαν χτίσει τα σπίτια τους, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνεια, με τα οποία κατασκεύασαν τις οικίες τους. Από 250, από 250 δάνεια που δόθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν όλα για να κτιστούν οικίες και ήταν πολύ καλά σπίτια και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ θετικό γιατί έχω δει και την άλλη πλευρά, τις χειρότερες εγκαταστάσεις τέρσης. και οι Ρωμά θεωρούσαν πολλοί από αυτούς ότι δεν χρειαζόταν να ξεπληρώσουν τα δάνεια, δεν ξεπληρώναν τα δάνεια αυτά και επομένως η ελήψη πληρωμών οι τράπεζες θέλησαν να ξαναπάνουν πίσω τα σπίτια. Υπήρξε λοιπόν μια σύγκρουση. Από τη μία μεριά έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο δίδει δάνεια τα οποία έχουν σαν στόχο τη στο Ρώμα και ένα άλλο Υπουργείο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει τις τράπεζες και να δώσει τα χρήματα στην τράπεζα για να καλύψει το κόστος των δανείων. Υπάρχει και πρόβλημα επίσης με τους ε, πιστωτές στο Ρωμά. Μπορεί να χωροστάνε μικροποσά. Για χίλια ευρώ, παραδείγματος χάρη, για να βάλουμε μια αντένα τηλεόραση στο σπίτι και μετά επειδή δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα ποσά αυτά έρχεται ο πιστωτής και ζητάει την κατάσχεση του σπιτιού. Αυτό το οποίο ζητούν λοιπόν που ζητούμε να γίνεται τώρα από την ε, κυβέρνηση είναι να υπάρξει κάποια μορφή συντονισμού. Να μην δίνουμε με το ένα χέρι και να παίρνουμε με το άλλο. Και να αλλάξουμε και την νομική βάση των προγραμμάτων ώστε να μπορούν να κάνουν μικρές πληρωμές οι Ρωμά σε πιο εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επιτυχία στα προγράμματα αυτά. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας τονίσω ότι εάν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης, αν υπάρχει στάση ευθύνη από την πλευρά των ατόμων και αν προσπαθείτε να βρείτε μηχανισμούς για να προσαρμόσετε τη λύση των προβλημάτων στις τοπικές ανάγκες μπορείτε να προέρχονται καλά αποτελέσματα σε άλλες περιοχές. Περιοχές που είναι πλήρως εγκατεστημένοι η Ρωμά και δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Ελλήνων Ρωμά και μη Ρωμά, το πρόβλημα είναι πολλές φορές να βρεθεί γη για τους καταβλισμούς τους, για να μπορέσουν να διευρύνουν τους καταβλισμούς τους. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά ε, ε, δημιουργίας καταβλισμών στο βορρά της ε, Ελλάδος σε μια περιοχή που λέγεται Δροσερό έξω από την Ξάνθη υπάρχει μια αφαίρετη πόλη των Ρωμά και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και για να νομιμοποιήσουν τη γη στην οποία έχουν χτίσει τα σπίτια τους και τα ίδια τα σπίτια τους. Εφόσον είναι αυθαίρετες κατοικίες λοιπόν πρέπει να τις νομιμοποιήσουν και επίσης πολλές φορές πρέπει να αλλάξουν την ε, μορφή των κατοικιών τους για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για υδροδότηση, ηλεκτροδότηση κτλ. Βλέπετε λοιπόν δεν μπορεί να έχει κανείς κανόνες in abstracto οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται στους Ρωμά. Θα πρέπει να υπάρχουν προσαρμογές σε εθνικό επίπεδο για τις ανάγκες τους. Τις περιοχές λοιπόν αυτές όπως της ε, Ξάνθης όπου υπάρχει παράνομος χαρακτήρας της κατοχής της γης και της οικοδόμησης ε, κατοικιών, θα πρέπει να υπάρξει κάποια κρατική παρέμβαση για να νομιμοποιηθούν αυτές οι οι εγκαταστάσεις και να μπορούν να έχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες ηλεκτροδότησης, ε, υδροδότησης, αποκομιδής απορριμμάτων, σχολεία και παιδική σταθμή, συγκοινωνιακές ε, γραμμές κτλ. Του τουλεχθέντος πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πολλοί Ρώμα που ζουν σε απόλυτα παράνομους καταφλισμούς που είναι αυτοσχέδιες που έχουν αυτοσχέδιες κατοικίες από πλαστικό, ξύλο, από γυαλοβάμβακα κτλ. Βέβαια, αυτές οι αυτοσχέδιες κατοικίες δεν τους δίνουν ουσιαστική προστασία από τα στοιχεία της φύσης και πολλές φορές είναι επικίνδυνες και για τη δική τους ζωή και διαβίωση. Γιατί στερούνται τρεχούμενο νερού, ηλεκτρισμού, ε, αποχωρητηρίων ή οποιοδήποτε υποδομών που θεωρούμε απαραίτητες για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι λοιπόν σε αυτούς τους χώρους που ζουν οι περισσότεροι μετανάστες ε, Ρωμά σε συνθήκες οι οποίες είναι πραγματικά ικτρές. Το να δημιουργηθούν οι βασικές υποδομές για αυτούς λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι τοπικές αρχές να αναλάβουν τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Στη χώρα μου οι τοπικές αρχές είναι υποχρεωμένες ε, νόμου να δημιουργούν ε, κατάλληλους για τους Ρωμά οι οποίοι διακινούνται για λόγους οικονομικούς, για λόγους επιβίωσης. Μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο λοιπόν οι εθνικές αρχές για την κατασκευή και την διαχείριση αυτών των καταβλισμών. Αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι αν αυτοί οι καταβλισμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μόνιμοι, θα μεταβληθούν σε εγκέτο. Γι' αυτό αν μιλάμε για μικρούς καταβλισμούς θα πρέπει να, βρουν, να βρεθούν άλλοι τρόποι από τις αρχές να αντιμετωπιστούν αυτοί οι καταβλισμοί και όχι με τη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων διαβίωσης. Αλλά όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί δεν υπάρχει άλλη λύση παρά οι καταβλισμοί οι οποίοι δημιουργούνται από τις τοπικές αρχές. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα όλοι αυτοί οι πληθυσμοί να έχουν ε, στέγαση. Σας παρακαλώ να συντομεύετε, λέγεται, λέει η πρόεδρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, είναι πολύ ενδιαφέροντα, δεν έχουμε χρόνο. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν τώρα είναι το εξής. για να αλλάξουμε τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι Ρώμα, θα πρέπει να υπάρξει και μια αλλαγή στην αντίληψη. Μιλήσαμε για, την, για το στιγματισμό, το Ρωμά, για τις διακρίσεις σε βάρος τους. Πιστεύω ότι ο ρατσισμός και η διάκριση αυξάνει όταν οι άνθρωποι θεωρούν ότι απειλούνται και ότι η ποιότητα ζωής τους απειλείται από την παρουσία των παρανόμων αυτών μεταναστών. Δεν ξυπνάει κανείς μια μέρα λέει δεν τους πάω και τους μισώ τους Ρωμά. Αυτή η εχθρότητα αρχίζει να εκφράζεται όταν θεωρεί κάποιος ότι κινδυνεύει η ζωή τους όταν υπάρχει ρήπανση από τις ε, φωτιές που ανάβουν, παραδείγματος χάρη, από τα σκουπίδια που πετάνε, όταν υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες. Αναφέρθηκε το θέμα της εγκληματικότητας. Οι Ρωμά δεν είναι εγκληματίες. Αν κάνουν, ε, κάνουν δραστηριότητες που είναι παράνομες, το κάνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εδώ εμπλέκεται και η ευθύνη του κράτους. Είναι απαραίτητο να ληφθεί αυτό υπόψη. Θα πρέπει να τροποποιήσει κανείς τις συνθήκες της πραγματικής ζωής και αν γίνει κάτι τέτοιο, όταν υπάρχουν επιπλέον διακρίσεις, τότε θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει κανείς. Αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσει κανείς μια κατάσταση η οποία τρέφει, εκτρέφει τη διάκριση καταρχήν. Και το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι η παιδεία. Δεν βλέπω κανένα τρόπο να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ρωμά παρά μόνο μέσω της παιδείας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε μια γυναίκα στο γραφείο μου η οποία δεν είχε καθόλου έγγραφα, δεν είχε υπηκότητα, δεν είχε καμία δυνατότητα να πάρει διάφορες παροχές. Εγώ άκουσα το παραπονό της και πήρα τηλέφωνα για να μπορέσει να πάει στο γιατρό γιατί ήταν άρρωστη και τα λοιπά. Την άλλη μέρα επανέρχεται στο γραφείο μου και ρώτησα τι έγινε, τι συνέβη. Και είχε τα δύο παιδιά της μαζί και ήρθε να μου παρουσιάσει την κατάσταση το πρόβλημα μιας άλλης γυναίκας. Το πρόβλημα που είπα είναι γιατί δεν τα παιδιά στο σχολείο. Είπε γιατί δεν έχουν χαρτιά. Και είπα, γιατί δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο παρά το γεγονό ότι δεν έχουν χαρτιά. Υπάρχει μια πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση ότι όλα τα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο ανεξάρτητα από το αν έχουν χαρτιά και άδειε διαμονή ή οτιδήποτε τέτοιο. Λέει, μα δεν έχουν τα ρούχα να πάνε στο σχολείο. Και τότε θύμωσα μαζί τη της είπα, θες τα παιδιά σου σε 10-20 χρόνια από τώρα να είναι στην ίδια κατάσταση που είσαι εσύ τώρα. Αν τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο, θα είναι στην ίδια κατάσταση. Πρέπει αύριο να πας να τα γράψεις στο σχολείο. Και είπε πάλι την επόμενη μέρα και είπε πήγα στο σχολείο. Και μου ζήτησε ο διευθυντής του σχολείου χαρτιά για τα παιδιά. Ένιωσα μεγάλη έκπληξη γιατί δεν φανταζόμουν ότι θα πάει στο σχολείο. Και πάλι χρειάζεται να παρέμβουμε και να πείσουμε το σχολείο να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Αλλά πιστεύω ότι όταν ξεκινάτε με μια πρωτοβουλία, όταν προσπαθείτε να πείσετε τους ανθρώπους να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής τους, θα το κάνουν. Το να μην επιτρέπεται στα παιδιά το Ρωμά να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, αυτό είναι ένα μεγαλύτερο έγκλημα από το να τα σκοτώνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την παιδεία των ε, παιδιών αυτών των Ρωμά. Ευχαριστώ. Thank really have... Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λυπούμε που αναγκαζώ να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να δούμε πόσο δύσκολο και πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα. Μιλούμε για στρατηγική πλαίσιο, αλλά τι σημαίνει, εδώ υπάρχουν τόσο συγκεκριμένα προβλήματα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή και στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτούς που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ιδιαιτέρως για τα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που δώσατε. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Πιερ Μπάρς να προχωρήσει στην ε, ε, παρουσίασή του και μετά θα έχουμε λίγο μόνο χρόνο για ε, συζήτηση. Ελπίζω ωστόσο κάπως να τα καταφέρουμε. Έχετε το λόγο. Είναι καλό ή κακό να μιλήσει κανείς τελευταίος. Σας ευχαριστώ πάντως εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπεράσπισης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και θυμίζω ότι η κακο να μιλησει κανεις τελευταιος σας ευχαριστω παντως εξ ονοματος της ευρωπαικης ενωσης Υπεράσπιση των ανθρωπινων δικαιωματων και θυμιζω οτι η οργανωση μας, στην οργάνωσή μας συμμετέχουν 25 οργανώσεις ε, ευρωπαϊκές. Θα προσπαθήσω να θυμίσω ορισμένα πράγματα, ίσως σε ένα διαφορετικό τόνο. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, έστω και αν θα μπορούσα να σας πω πολλές. Θα θυμίσω μόνο ότι τα γεγονότα του θέρους 2010 στην Γαλλία είναι ε, σημάδια μιας, δυστυχ... μιας ατυχούς πολιτικής που στιγματίζουν ένα, ε, μια πληθυσμιακή ομάδα, τους ε, Ρώμα, που είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι και με τον τρόπο αυτό έχουν τα ίδια δικαιώματα όπω όλοι οι Ευρωπαίοι υπηκοί και επομένω και την προστασία από πλευρά των ε, δημοσίων ε, ε, υπηρεσιών. Οι περισσότεροι από αυτού είναι φτωχοί άνθρωποι και οι κυβερνήσει του κάνουν συχνά από τράγου τράγους των οικονομικών δυσχεριών. Συχνά περιθωριοποιούνται, συχνά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν άμυνε και είναι θύματα τελικά ενό πολιτικού λόγου θέματα ασφάλειας που τους βάζουν μαζί με την, ε, στο ίδιο επίπεδο με την τρομοκρατία. Μιλούμε για πορτοφολάδες στην πραγματικότητα. Μέχρι εκεί είναι η ε, εγκληματική του δραστηριότητα. Εφόσον τους δίνεται η δυνατότητα, εγκαθίστανται σε δημόσια ε, εδάφη και θέλουν μετά να τους διώξουν για να ικανοποιήσουν τις πιέσεις από τα αστικά κέντρα. Τους ζητούν να μην είναι πλέον ορατοί, να εξαφανιστούν ως λαός. Το φαινόμενο αυτό δυστυχώς δεν είναι νέο και δείχνει τα όσα έχουν συμβεί και παλαιότερα και στο 19ο και στον 20ο αιώνα και μάλιστα ήταν και θύματα γενοκτονίας στο ναζιστικό καθεστώς. Σε μια λογική αποκλεισμού, ξενοφοβίας, συνολικού χαρακτηρισμού που τους ε, κάνουν στην πραγματικότητα να είναι, όπως είπα, ε, τα θύματα από τα προβλήματα της ε, κοινωνίας με την ανεργία και ούτω καθεξής. Αυτά που συνέβησαν στη Γαλλία το προηγούμενο καλοκαίρι δεν είναι μοναδικά στην Ευρώπη. Τους έβαλαν όλους μαζί τους ανθρώπους αυτούς για παράδειγμα, και ήταν, ενώ ήταν και Βούλγαροι υπήκοοι και Ρουμάνοι υπήκοοι κλπ. Οι τόποι κατοικία του καταστράφηκαν τα τροχόσπιτά τους και ούτε καθεξή. Επανελήφθηκαν τέτοια σενάρια όπω και σε άλλε χώρε, όπω το 2007 στην Ιταλία, με οδήγησε στο θάνατο μια γυναίκα, στην καταστροφή των στρατοπέδων, στην απέλαση των ε, Ρώμα ακόμα χειρότερα. Μετά τα όσα έγιναν στη Γαλλία, ο, το Ιταλός υπουργό επανήλθε και και το 2005 στην ε, Πάτρα ε, εκδιώχθηκαν από τους καταβλισμούς τους ε, οι Ρώμα. Όλα αυτά γίνονται συνήθως ε, μέσω των αστυνομικών αρχείων, τα οποία πολλαπλασιάζονται και μας ανησυχεί αυτό ιδιαίτερα. Θα πρέπει να καταδικαστεί έντονα. Ανάμεσα σε άλλα γεγονότα, η Γερμανία αυτή τη στιγμή στέλνει πίσω τις οικογένειες ε, Ρώμα στο Κωσυφοπέδιο, που έχουν έρθει στο, στη Γερμανία, έχουν μεορφωθεί στα γερμανικά και έχουν ζήσει στην Γερμανία, έχουν μεγαλώσει μάλλον στη Γερμανία. Είτε είναι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Σκοτία, στην Ουγγαρία, οπουδήποτε η κατάσταση είναι η ίδια. Οι Ρωμά ορίζονται ως χωριστή κοινωνική ομάδα με ομοιογενή χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, τον τόπο κατοικίας τους και τον τρόπο ζωής τους. Είναι κάτι το οποίο, μια εικόνα η οποία διατηρείται και από τις πολιτικές αρχές με βάση ιστορικοκοινωνικά χαρακτηριστικά και με βάση την ε, κινητικότητά τους ή το αντίθετο, η κατάστασή τους είναι ξεχωριστή στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εάν δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε τι ακριβώς είναι η Ρώμα, μόνο οι ίδιοι μπορούν να το δηλώσουν, να το πούνε, να πούνε ότι θέλουν να ζουν με τον τρόπο, έχουν το δικαίωμα να ζουν με τον τρόπο τον οποίο έχουν επιλέξει και μέσα σε έναν κόσμο όπου οι διαφορές ε, ε, αναγνωρίζονται και όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει όπως ε, θέλει, θα πρέπει και οι Ρώμα να μπορούν να, να, να, να κάνουν το ίδιο. Συχνά όμως είναι ανεπιθύμετοι ε, συχνά θα ήθελα να είναι αόρατοι, τα δικαιώματά τους παραβιάζονται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμβάσεις και τις ε, αρχές που ορίζονται στις συνθήκες της ε, ε, ΟΚ. παρά την απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πρόεδρος ζητά από τον ομιλητή να μιλήσει λίγο πιο σιγά για να τον προλαβαίνουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν Παρά λοιπόν τις ε, εκθέσεις και τις ε, γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου, σε αντίθεση με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει ενταχθεί στι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ρωμά εξακολουθούν να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και θα κάνω κάποιε παραθέσει ε, από αυτόν τον χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη και πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται. Κάθε πολίτης τη Ευρωπαϊκή ένωση έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην, ε, στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής, τη οικογένεια του. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ε, εκπαίδευση και στην εργασία. Οι, οι συλλογικές απαγορεύονται απαγορεύεται κάθε διάκριση. Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Η προστασία της ε, οικογένειας ε, ε, ισχύει στο δικαστικό, κοινωνικό και πλαίσιο. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην υγεία και ένα χέρι υγειονομική περίθαλψη. Κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα να εισακουστεί πριν να το απαγγελθεί καταγγελία. Υπάρχει υποχρέωση για την διοίκηση να προστατεύει αυτά τα δικαιώματα και κάθε άνθρωπο του οποίου τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να είναι εγγυωμένα και όλα ε, και για αυτούς που ορίζονται ως Ρωμά. Ας θυμηθούμε τον Σπίτλα το 2007, τον Επίτροπο, σε σχέση με τα όσα έγιναν στην Ιταλία. Και που δεν ήταν μια μεμονωμένη υπόθεση. Η ρατσιστική βία τρέφεται από το λαϊκισμό, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε σε διάφορα κράτη-μέλη. Ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεπεράσει το ρατσιστικό μίσος και την καταστρο... τα απογκρόμια και την καταστροφή μέσω της φωτιάς. Πώς ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά ενώ η κοινωνία δεν μπορεί να τους δώσει την ε, υγειονομική περίθελψη την κοινωνική βοήθεια αλλά ούτε και την ε, κατάλληλη εκπαίδευση. Πώς να, να μην αναφερθούμε στα ειδικά σχολεία και την αναγκαστική τους, ε, τον αναγκαστικό τους εκκλεισμό. Πώς να μην αναφερθούμε στα τέλη του μόλις του 20ου αιώνα την, τον αποκλεισμό των Ρωμά. Τέτοιες πρακτικές ακόμα ακολουθούνται. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε άγρυπνοι. Η εξαφάνιση ενός τέτοιου λαού θα είχε συνέπειες. Αν θέλουμε να... Εάν δεν αντιδράσουμε, τότε η ανθρωπιά μας θα εξαφανιστεί εκτός από αυτό το λαό και θα προχωρήσουμε προς το χειρότερο. Θα πρέπει λοιπόν, πέρα από τις ε, διασκέψεις και τις διάφορες εκθέσεις των ΜΚΟ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πέρα από την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων που μόλις σας ανέφερα, καταρχήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πραγματική χρήση των χιλιάδων ευρώ που προβλέπονται για αυτά τα, για αυτά τα προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω του εντοπισμού των συγκεκριμένων τελικών δικαιούχων, να απαιτήσουμε τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά και ε, τη διαφάνεια των δικαιούχων και των ΜΚΙΟ. Δεν χρειάζεται τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, θα μπορούσα βέβαια να επεκταθώ. Ε, υπηρεσίες ποιοτικέ που θα αντιστοιχούν σε αυτές που μπορούν να, τον οποίο μπορούν να χαίρουν και άλλοι πολίτες. Εάν συμφωνούμε πως όλες οι αποφάσεις εφαρμοστικές θα πρέπει να λαμβάνονται όσο γίνεται πιο κοντά στον δικαιούχο, τι θα συμβεί όταν δεν γίνεται τίποτα, τι θα γίνεται όταν οι τοπικές αρχές στη Γαλλία ή στην Αγγλία και σε άλλες χώρες θα πρέπει να δώσουν ε, εδάφη, να δώσουν χώρους γη στους, όσους, στους ταξιδιώτες που αποφασίζουν να εγκατασταθούν κάπου και δεν γίνεται τίποτα ε, θα πρέπει να μπορούμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Αυτό σημαίνει σε περίπτωση όπου οι τοπικές αρχές, οι κρατικές αρχές δεν εφαρμόζουν μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, να μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια, σε περίπτωση δηλαδή που οι τοπικές ή οι κρατικές αρχές δεν, προβαίνουν δεν ασκούν τα καθήκοντά τους. Και νομίζω πως αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση έχουμε πέσει. Και δεν επανέρχομαι στο θέμα της διαμεσολάβησης, το οποίο εξαιρετικά αναφέρθηκε η συνάδελφος. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην δικαιοσύνη ε, αυτό σημαίνει το δικαίωμα προσφυγής για κάθε άνθρωπο που αισθάνεται ότι, δεν, ότι, δεν, ότι καταπατώνται τα δικαιώματά του θα πρέπει τα εν λόγω άτομα να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, πράγμα που απαιτεί την ε, δημιουργία, απαιτεί μάλλον την δημιουργία κατάλληλων μέσων για την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Είναι παράδοξο τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει στόχο την κινητικότητα των πολιτών και θα πρέπει να σα πω ότι τις τελευταίες μέρες υπό την Βελγική Προεδρία παρακολούσα διάφορα συνέδρια, σεμινάρια που γίνεται λόγο για την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών εντό τη Ένωση, Μα όταν διακηρύσουμε τέτοιου επίσημού στόχου, η κινητικότητα των ανθρώπων που είναι πιο ευάλωτοι και πιο φτωχή, ε, ταυτόχρονα καταστέλλεται, αυτό δεν είναι αποδεκτό. 10.000 με 15.000 άνθρωποι, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν σε μια χώρα που δεν είναι δική τους και που περιλαμβάνει 65 εκατομμύρια ανθρώπου και να λέει κανείς ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κινδυνεύει να κάψει ολόκληρη τη χώρα δείτε ποιο είναι το ποσοστό αυτών των ανθρώπων θα δείτε ότι είναι απειροελάχιστο και τέλος δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε μάλλον τα ποσοστά στην επίτευξη των στόχων, να, να, να κερδίσουμε, να νικήσουμε έναντι της φτώχεια και του αποκλεισμού, δεν είναι θέμα ποσοστών, είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα. Θα πρέπει να ληφθούν ε, τα απαραίτητα μέτρα ώστε 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες να βγουν από τη φτώχεια και από τον αποκλεισμό στον οποίο έχουν περιοριστεί. Ε, να μπορούν να βρίσκονται σε ισότιμου όρου με τους υπόλοιπου Ευρωπαίους πολίτες και να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. Ευχαριστώ. Thank you very much for your... Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ομιλία σας. <clears throat> Είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί κιόλα ότι και όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας λόγω της οικονομικής κρίσης πλήττουν τους πιο ασθενείς, εν προκειμένου τους Ρώμα. Ήταν νομίζω πολύ σημαντική αυτή η τελευταία σας παρουσίαση σε όλη την ακρόαση. Τώρα βέβαια ο χρόνος που μας μένει είναι πολύ περιορισμένος για να ακούσουμε ωστόσο μερικές παρεμβάσεις, ερωτήσεις, σκέψεις και μετά θα παρακαλέσω τους πανελίστ να ε, απαντήσουν. Η Λίβια πρώτη, χωρίς μικρόφωνο. Μετά από ό,τι ξέρω ο κ. Ιωάννης Βέντενικ της UNICEF θέλει να απευθυνθεί στο πάνελ. Σημειώνουμε εδώ τα ονόματα βέβαια. Παρακαλώ να είστε βέβαια σύντομες και σύντομοι διότι χάνουμε την ώρα, δηλαδή περνάει ο χρόνος μας και δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Η Λίβια. Δεν μίλησα πριν γιατί έχω την τάση να μιλώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω τη Γιονάρση για τη δική σας δηλαδή παρέμβαση γιατί ακούσαμε πράγματα από αυτά που είπατε από την, προοπτική, από την οπτική σας δηλαδή. Ε, αυτά θέλαμε να ακούσουμε από όλους τους ομιλητές, δηλαδή ποια είναι η δική τους οπτική γωνιά. Βέβαια ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά πρέπει να δράσουμε με επαγγελματικό τρόπο, όπως ε, πράττει η δική σας ε, οργάνωση. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ, διότι σπανίως βλέπω εθνικούς αξιωματούχους που να κατανοούν το θέμα τόσο καλά όσο εσείς και που ε, δρούν χωρίς ε, τέτοια ε, gypsy business. Δεν σας έχουμε ξαναδεί σε άλλη διεθνή συνάντηση. Θα θέλαμε πολύ να έχουμε τις πληροφορίες αυτές, το feedback αυτό που δίνετε από την καθημερινή εργασία σας. <coughs> βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα τέλος εσά κύριε ε, να σας ε, υποβάλω ένα ερώτημα. Είπατε ότι ακόμα και αν μέτρα λαμβάνονται και απέναντι στις αρχές ή τουλάχιστον αν ζητείτε από τις αρχές, αν ζητούνται από τις αρχές να, λαμβάνουν, να λάβουν μέτρα, λίγα πράγματα γίνονται. Ποια μέτρα έχουν ζητηθεί από τις ε, γαλλικές αρχές, από την ε, ε, Ομοσπονδία σας, γιατί δεν είναι μόνο οι Βούλγαροι και ε, Ρουμάνοι Ρώμα που εφήγησαν από τις ε, δράσεις αυτές, αλλά και ήδη οι Γάλλοι. Τώρα, για, αυτά, για αυτούς τους παρόνομους καταβλισμούς στην Ιταλία, Ελλάδα ή Γαλλία. Από τους Ρώμα το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι μόνο οι γιατροί χωρίς σύνορα τους επισκέφτονται καθημερινά και τους βοηθούν καθημερινά. Δεν έχω ακούσει ποτέ για οργάνωση Ρώμα ή μη Ρώμα που πήγε στους ανθρώπους αυτούς, στους καταβλισμούς αυτούς, οι οποίοι έρχονται ε, από, σαν, σαν να είναι από το πουθενά, δεν έχουν που να μείνουν, δεν έχουν απολύτως τίποτα, καμία πληροφορία και πάνε και εγκαθίστανται σε κάποιο καταβλισμό. Σπανίως, σπανιότατα ακούω από τις ε, ε, οργανώσεις αυτές πώς βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς. Εδώ μιλούμε τόσο πολύ για την ευαισθητοποίηση. Ναι, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και πολύ άσχημη από την πλευρά των μίδια Πώς είναι δυνατόν όλες αυτές οι οργανώσεις να μην προσπαθούν να μιλήσουν για τον ρόλο των μίδια, των μέσων. Γιατί η καλύτερη ε, εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα ήταν εάν αυτά τα μέσα ενημέρωσης για τα οποία όλοι πληρώνουμε ως Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και θα έπρεπε να είναι αντικειμενικά. Θα έπρεπε να επιμείνουμε εμεί ως Ευρωπαίοι πολίτες να δίνουν τα μέσα αυτά μια αντικειμενική εικόνα των Ρώμα. Δεν με ενδιαφέρει μια ε, εκστρατεία που να λέει τι καλή που είναι η μη Ρώμα ή όσοι δεν είναι Ρώμα. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, ο ρόλο των ε, μέσων θα έπρεπε, είναι τεράστιο εδώ, εν προκειμένου. Και όχι να ε, προωθούν μια εντελώ παράλογη ιστερία. Καλύτερα να ακουστούν οι φωνές των ίδιων των ανθρώπων. Και να μην πολιτικοποιείται το θέμα, ούτε, όπως είπα, να καταλήγει σε μια ιστερία. Αυτά ήθελα να πω. Το ερώτημά μου είναι τι είδους μέτρα ζητήσατε ε, ε, από τις γαλλικές αρχές για τους ταξιδιώτες αυτούς. κυρία Ακολουθεί η κυρία Φλότρο και ο κύριο Βέντενινγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργηθεί τον, ε, το Μάρτιο να είναι σωστά βασισμένο για μια στρατηγική περιεκτική και για να ευδοκιμήσει θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον αγώνα κατά των διακρίσεων και στο νομικό επίπεδο σε αποτελεσματικό επίπεδο. Παράδειγμα της Γαλλίας. Μου είπε κάποιος ο οποίος τα για τρία χρόνια ε, διευθυντής αστυνομίας της νομαρχίας του Παρισιού είπε ότι έχουμε κάποιους περιορισμούς αλλά έχουμε ποσοστώσεις για τις εκδιώξεις. Όταν έρχεται λοιπόν ο Σεπτέμβριος και δεν έχουμε συμπληρώσει την ποσόστοσή μας, τι κάνουμε, βρίσκουμε τους Ρωμά και τους διώχνουμε. Και δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούν πολύ γιατί ξέρουν ότι θα ξαναγυρίσουν, δέχονται να φύγουν ε, θελοντικά να τους δώσουμε 200-300 ευρώ γιατί δεν τους κοστίζει πολύ και το ταξίδι πολύ πιο εύκολα να του διώξουμε αυτού παρά να διώξουμε Ασιάτε ή κάποιου άλλου. Λοιπόν, σα το δίνω αυτό σαν παράδειγμα. Την άνοιξη θα πούμε στη Γαλλία, σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αναπτύξτε μια εθνική στρατηγική για την ενσωμάτωση των Ρώμα. Αλλά συγχρόνω υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά η οποία είναι απόλυτα διακριτική συνεχιστή στη Γαλλία ή και σε άλλες χώρες, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βασιστούμε και στον αγώνα κατά της διάκρισης. Και υπάρχει και μια δυσκολία όταν οι κυβερνήσεις αντιτίθενται ουσιαστικά, αδρανούν και χρονοτριβούν για να πάρουν μέτρα για την ενσωμάτωση των ε, Ρωμά, γιατί τους βολεύει να τους έχουν σαν αποδιπομπέους τράγους σε πολιτικά αντικό επίπεδο θα πρέπει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο άμεσα παρακάμπτοντας τα κράτη να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές γιατί στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλές τοπικές αρχές που κάνουν καταπληκτικά πράγματα για να βοηθήσουν τους, Ρώμ, τους Ρώμα αλλά αν δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από την εθνική κυβέρνηση για να πάρουν αυτά τα κονδύλια είναι πολύ δύσκολο ο ρόλο του, είναι πολύ δύσκολο το έργο του. Πιστεύω τέλο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνδυάσει τι δράσει τη με τι δράσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη γιατί εγώ είχα οργανώσει μια συνάντηση με τους Ρωμά από την Ισπανία, την ε, Ιταλία και τόνισαν όλοι ότι είναι απαραίτητο, είναι κέριο το να υπάρχουν μεσολαβητές για τους Ρωμά οι οποίοι μπορούν να είναι συνομιλητές τους με τα σχολεία, με τις δημόσιες αρχές κτλ. Αν έχετε ένα πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή η εκπαίδευση των, ε, και η απασχόληση μεσολαβητών όπως τους εκπαιδεύει και τους ε, χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για μένα αυτό είναι κεφαλαιόδης. Just one Κύριος Βέντελινγκ και μετά θα ήθελα να ζητήσω από το πάνελ να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Κύριος Βέντελινγκ καταρχήν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η εκπαίδευση είναι το πιο βασικό στοιχείο για σώμα, αλλά θα έλεγα ότι η νεαρή ηλικία και η ανάπτυξη των γνώσεων στην ε, προσχολική ηλικία τα πρώτα τρία χρόνια, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Ό,τι χάνει ένα παιδί τα πρώτα τρία χρόνια δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Αυτό σημαίνει εκπαίδευση και τον... Ε, γονέων στο επίπεδο πριν από τη γέννηση του παιδιού και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και μεγαλύτερες γλωσσικές διευκολύνσεις για αυτόν τον πληθυσμό πρέπει να είναι ένας από τους κύριους πυλώνες οποιασδήποτε στρατηγικής ή παιδική και νηπιακή ηλικία. Ένα άλλο στοιχείο είναι η επίπτωση του καθεστώτος υπηκότητος για το καθεστώς στο οποίο βρισκόνται τα παιδιά αυτά. Βλέπετε ότι αν επισφαλίσει η κατάσταση των παιδιών, αυτό ουσιαστικά αποτρέπει τα παιδιά από το να εποφεληθούν από το σχολείο. Οι προσπάθειέ τους πηγαίνουν στράφη σε αυτές τι περιπτώσεις. Επομένω, το καθεστώ των παιδιών αυτών έχει άμεση επίπτωση στην παιδεία τους και επίσης υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούμε να τι λάβουμε υπόψη, όπως είναι το λεγόμενο coaching, η υποστήριξη αυτού του είδους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους Ρωμά από τον, μέσα στις κοινωνίες μας και επίσης η αναθεώρηση της οδηγίας επιστροφής του 2008 και το να διασαφινιστεί τι είναι ακριβώς το καλύτερο συμφέρον του παιδιού σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο ε, αναπαραγωγής της ένδυας από μία γενιά στην επόμενη. Κύριε Ντεμιρόσκη, σε πέντε λεπτά πρέπει να φύγουν διερμηνείς. Παρακαλώ να είσαστε σύντομος. Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή αυτή η άσκηση, αυτή η ακρόαση για το τι θα πρέπει να περιέχει σε επίπεδο διανοητικό και ενοιολογικό η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης να εξελθεί από αυτή την ακρόαση είναι ότι εσείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έρθετε πιο κοντά στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει μια διαφορετική θέση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς μικρόφωνο κυρία Γιάρουκα. Όχι, η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ σαφή και πάρα πολύ ειλικρινή. Ο κύριο Άντορ ήταν πολύ ειλικρινή. Είπε ότι το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στη δράση των κρατών μελών, γιατί η ευθύνη βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Εμεί θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε να ξέρουμε ποιο είναι αυτό ο οποίο έχει εντολή για την εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Πάλι κυρία Γιάρουκα χωρί μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι λέει. Θα μην υπάρξει λοιπόν σύγχυση και παρεξήγηση για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και πού βρισκόμαστε. Έχουμε μία πολιτική υποστήριξη από το Κοινοβούλιο μια θέση του Κοινοβουλίου και μια θέση της Κομισιόν. Αυτές οι δύο θέσεις θα πρέπει να συγκλίνουν. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η γαλλική κυβέρνηση διατυπώνει ένα κείμενο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρωμά. Μήπως πρέπει να το συζητήσουμε και με τους Γάλλους. Μήπως πρέπει να καλέσουμε και άλλα κράτη-μέλη να μας δώσουν τις απόψεις τους. Πρέπει όλοι να δώσουν την άποψή τους για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευχαριστώ. σίγουρα. Νομίζω αυτό είναι, το είναι ένα πρόβλημα, γιατί προσπαθούμε ακριβώς να διευρύνουμε τη δημόσια ακρόαση γιατί έχουμε πολλά εκκρεμή ερωτήματα. Δεν είναι το τέλος αυτή εδώ η ακρόαση. Ακούσαμε θέσεις, δηλώσει από όλες τις πλευρές. Ε, πραγματικά θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις κοινότητες, με τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. Πάντως και για σήμερα ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Μπορούμε σίγουρα να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε την, την, την συζήτηση αυτή. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα τρία λεπτά για να δώσουμε το λόγο στους μιλητές μας για να κάνουν κάποια πολύ σύντομα σχόλια. Καταρχήν η Ιζαμπέλ χαλάσει Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θα αναφερθώ στο τελευταίο στη τελευταία παρατήρηση, γιατί και η Λίβια αναφέρθηκε σε αυτό. Η Κομισιόν έχει υποβάλει προτάσεις και το, αυτό που θέλουν είναι να καλέσουν τα κράτη-μέλη να φτιάξουν στρατηγικές, να τις ε, μεταρρυθμίσουν με βάση κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Και είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το πάρει αυτό σοβαρά υπόψη και να το αντιμετωπίσει σε άμεση συνεννόηση με την Κομισιόν και να ζητήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, μια στρατηγική της της Κομισιόν. Όπου θα τοποθετηθεί στη θέση του συντονιστή για τις εθνικές στρατηγικές που θα απαιτηθούν από τα κράτη-μέλη. Γιατί διαφορετικά φοβάμαι ότι θα υπάρξει ένα κενό και θα χαθεί αυτή η διαδικασία, η ευκαιρία. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Ε, Επίση, πιστεύω πως ε, η διαδικασία θα πρέπει να αφορά τους δύο πυλώνες, κοινωνική ένταξη αλλά και καταπολέμηση των διακρίσεων, πρόθεση, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα περισσότερα ζητήματα που προέκυψαν τελευταία σχετίζονταν με την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και είδαμε ισχυρές κυβερνήσεις με πολύ ισχυρές δημοκρατίες που τελικά εγκαταλείπουν, απογοητεύουν τους πολίτες τους όσον αφορά τις παραβιάσει αυτές κατά το Ρώμα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να πω περισσότερα. Πολύ θα ήθελα να απαντήσω μεμονωμένα σε κάθε μια από τις ερωτήσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα ρίξω τους συναδέλφους αν το κάνω αυτό. Ε, I ναι, Παπαδοπούλου, εγώ θέλω να πω ότι η θυματοποίηση και αποκλεισμό των Ρώμα δεν μπορεί να σταματήσει μόνο αν οι άλλοι κάνουν ε, την προσπάθεια ή αν τους δίνουν ε, δώρα, χρήματα, τους προσφέρουν ε, διάφορα. Οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουν ε, δράση, να είναι υπεύθυνοι σε όλες τις πτυχές της ζωής της οικονομία, ε, όσον αφορά δηλαδή την απασχόληση, την παιδεία, θα πρέπει οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν ενεργά, γιατί διαφορετικά ό,τι και αν έρθει από αλλού θα είναι πατεναλιστικό και θα συνεχίζει τον αποκλεισμό και την θυματοποίησή τους. Ευχαριστώ. Ναι ή αν χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό ύφο. Αυτό δεν είναι γιατί δεν συμμερίζομαι πολλά από αυτά που ελέγχθηκαν και ιδίω και την τελευταία παρέμβαση και τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ένα πολιτικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Έρχομαι, ήμουν πρόσφατα στην, στη Βουλγαρία, όπου ζήτησαν να υπογράψουν μία ε, αναφορά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόγραμμα τηλεόραση οι Ρωμά. Υπάρχει μια εκστρατεία τη άκρα δεξιά κατά τον Ρωμά. Όλα αυτά επιτρέπονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια οργάνωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως εγώ δεν μπορεί παρά να ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική τάξη σήμερα αντιμετωπίζει το θέμα το Ρωμά. Αν συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, θα φτάσουμε σε πράγματα που θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτό το ύφο σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμερίζομαι τις απόψεις που διατυπώσατε εδώ. Αλλά έχουμε και την πίεση του χρόνου. Θέλω να απαντήσω λοιπόν και να πω ότι εγώ δεν μιλάω εξ ονόμα της Γαλλικής Λίγας ή άλλων φορέων. Γιατί εμείς είμαστε οργανώσεις που δουλεύουμε επιτοπίως. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Λίγα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Γαλλία ήταν πάντα παρούσα μπροστά μαζί με τους Ρώμα στις ε, εκδιώξεις με δικηγόρους στα δικαστήρια και όλα αυτά. Και επιμένω στην ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα νομικής προσφυγής, γιατί τα άτομα αυτά πολλές φορές είναι τα πιο φτωχά και δεν έχουν τη δυνατότητα μόνοι τους να καταθέσουν αγωγές. Όταν τους, βάζουμε στα όταν τους στα λεωφορεία, χωρίς να τους ρωτήσουν, τους παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, τους ε, του φακελώναν, του διώχναν και τους λέγανε δεν έχετε το δικαίωμα να επανέλθουν. Και τώρα έχουμε βιομετρικού φακέλου για εσά και άμα γυρίσετε θα σα πιάσουμε αμέσω. Μήπω δεν πρέπει να γίνει κάτι στο επίπεδο αυτό. Προφανώ πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα για την παιδεία, για την εκπαίδευση και όλα αυτά τα πράγματα, όπω είπατε. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα και σε ένα πολιτικό επίπεδο, να καταγγείλουμε τι πράξει αυτέ, οι οποίε είναι απαράδεκτε, οι οποίε έχουν γίνει εναντίον ατόμων που απλώς χρησιμοποιείται το πρόσημα ότι είναι Ρωμά, ενώ πάρα πολλοί από αυτούς δεν ήταν Ρωμά και εναπόκειται όπως είπατε στους Ρωμά να πούνε ποιοι είναι και τι θέλουν, αλλά εμεί σε λίγα προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέλουμε να υπερασπιστούμε παντού τα δικαιώματα των ανθρώπων όταν καταπατούνται και αυτή τη στιγμή καταπατούνται πράγματι με τρόπο ιδιαίτερα πρόδειλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ήταν μια πολύ καλή σύνοψη λοιπόν. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν προσπάθειες και στον τομέα αυτό. Γιατί βλέπουμε τις κινήσεις των ε, τις ακροδεξιές κινήσεις, την προσπάθεια δημιουργίας μισαλοδοξίας και τους κινδύνους αυτούς. Από την άλλη πλευρά αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Λίβια έχεις, χωρίς μικρόφωνο Λίβια. Ήθελα να έχω μια απάντηση στο ερώτημά μου. Τι μέτρα προτείνεται για τη γαλλική κυβέρνηση. Τι θα χρειαζόταν η λεγόμενη Jean με μετακινούμενοι, πληθ, πληθυσμοί. Τι προτάσεις μπορείτε να κάνετε στην κυβέρνηση για να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Θα ήθελα να ξέρω ποια ήταν η προτάσή σας για αυτό το θέμα. Πρωτού ζητήσουμε μια απάντηση, θα ήθελα να ζητήσω από τους διερμηνείς αν μπορούν να δώσουν Ένα λεπτό, τρία σημεία μοναχα, τα πιο σημαντικά σημεία. Ωραία, παρακαλώ, αν μπορείτε. Θέλω ε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματο όλη τη ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γαλλία. Αλλά το θέμα αυτό στη Γαλλία, όπω και σε άλλε χώρε. είναι το εξή. Έχετε του λεγόμενου Σόντι του τους ε, Ρωμά, οι οποίοι είναι γαλλική υπηκότητα. Έχετε όμω και πληθυσμού στη Γαλλία που έχουν έρθει από άλλε χώρε. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν θα είναι διαφορετικά ανάλογα με την υπηκότητα, με την εθνικότητα αυτών των ατόμων η γαλλική κυβέρνηση. η Jean Voyage, όπως ξέρετε, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί είναι Ρωμά, αλλά δεν είναι όλοι αποκλειστικά Ρωμά. Ένα άτομο στη Γαλλία που έχει το χαρακτήρα του μετακινούμενου δεν μπορεί να πάει στην, ε, να πάει στην, ε, σε ένα σούπερ μάρκετ και να γράψει μια επιταγή γιατί έχει μονάχα την κάρτα του μετακινούμενου, αλλά δεν έχει μια μόνιμη άδεια διαμονής. Υπάρχει, υπάρχει λοιπόν υποχρέωση να εξωθούν αυτές οι καταστάσεις και θέλω να υπενθυμίσω ε, κυρία Φλότρο ότι υπάρχει μια οργάνωση η οποία αγωνίζεται διακόπτη πρόεδρος νομίζω ότι τώρα πρέπει να σταματήσω το επίσημο τμήμα της ε, συνεδρίασης Μπορείτε οι τρεις σας να συνεχίσετε αυτή τη συζήτηση και είμαι σίγουροι ότι είναι διαθέσιμη ακόμα η αίθουσα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να συνεχίσουμε οι διερμηνείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρία σε αυτή την πρωινή. Συνεχίστε και θα θέλαμε να ακούσουμε και τα πορίσματα των συζητήσεων σας.